Ξεκινάμε λοιπόν. Επαναλαμβάνω ότι η συνεδρίασή μα θα αναμεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν χθε στη συνάντηση των συντονιστών, χθες το βράδυ. Θα ζητήσουμε τη δυνατότητα έκθεσης πρωτοβουλίες για τους προσανατολισμούς για πιθανή μεταρρύθμιση των συνθήκων στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συναντηθώ και με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ για να συζητήσουμε τους τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στις δύο επιτροπές και πιθανώς να υπάρξει και μία μεικτή συνάντηση των συντονιστών των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αποφασίστηκε επίσης ότι η συγητής για την πρωτοβουλία των πολιτών θα οριστεί από την σοσιαλιστική ομάδα. Αλλά για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ο εισηγητής θα είναι ο συνάδελφος Μέσερ Σμιτ. Ζητήσαμε επίσης και μία μελέτη για τον δημοκρατικό έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στις συναντήσεις κορυφής. Τέλος, και σχετικά με τις επιτροπές έρευνας, εδώ δεν έχουμε τον συνάδελφο κύριο Μάρτιν που ασχολείται με το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να προσκαλέσουμε τον Προεδρείο και το Συμβουλίο στη συνάντησή μας της 20 Δεκεμβρίου για να ακούσουμε τις απόψεις του Συμβουλίου για τις εκθέσεις μας ή εάν η συζήτηση θα πρέπει να γίνει και η συνάντηση τον μήνα Ιούνιο. Αλλά αυτά θα μας τα πει ο Μάρτιν που θα έρθει αργότερα. Ένα συνάδελφος έχει ζητήσει το λόγο, ο κύριος Γκουερέρο. Ναι, ήθελα να σας πω ότι ο Ντέιβιτ Μάρτιν θα φτάσει λίγο αργότερα και θα μπορέσουμε να το ρωτήσουμε τότε για ποιο συγκεκριμένο λόγο θεωρεί σκόπιμο να ε, καλέσουμε την Πολωνική Προεδρία. Ε, Κύριε Μέντες πήγω. Πρόεδρε, για να διευκρινίσω κάτι που εχθέ ίσως δεν εξήγησα σωστά. Είμαι υπέρ της έλευσης της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Μου το ζήτησε ο κύριος Μάρτιν και είναι καλό. Αλλά δεν, δεν είμαι βέβαιος και λένε και άλλοι συνάδελφοι ότι είναι κατάλληλη ημερομηνία. Εχθές είπα ε, να ακούσουμε τον Ντέιβιτ, αλλά η ημερομηνία δεν ήταν ίσως η καλύτερη. Μου φαίνεται θετικό να έρθει η Πολωνική Προεδρία, αλλά να δούμε πότε. Α, και κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε, χτες στους συντονιστές μετά από αίτημα του κυρίου Νταφ προβληματιστήκαμε ε, αν θα ψηφίσουμε ή όχι τη γνωμοδότηση της κυρίας Ρέγνερ σήμερα. Πρέπει να το αποφασίσουμε και αυτό. Για την έκθεση, για την γνωμοδότηση μάλλον Ρέγνερ, αποφασίσαμε να ακούσουμε την άποψη της εισηγήτριας. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Πριν την ψηφοφορία όμως θα της δώσουμε το λόγο τίθεται το θέμα ε, γιατί ο κύριος Νταφ ε, είχε ζητήσει και την αναβολή αν ε, θυμίστε. Το θέμα είναι ότι η νομική επιτροπή δεν έχει ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα και αν μεταθέσει την απόφαση, την λήψη, την ημερομηνία λήψης της απόφασης, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Περιμένουμε και μία γνωμοδότηση λοιπόν για το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε ότι η Νομική Επιτροπή έχει αλλάξει τις προθεσμίες και έτσι αν δεν εκφράσουμε τη γνωμοδότησή μας σήμερα τότε έχουμε μείνει πίσω. Ο κύριος Γκερέρο, κοιτάξτε πρόεδρε, ευχαριστώ. Εχθές συμφωνήσαμε να περιμένουμε να έρθει η κυρία Ρέγνερ και να της πούμε ότι δεν θα ψηφίσουμε σήμερα, μάλλον να ζητήσουμε να αναβληθεί η ψηφοφορία για να μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη απάντηση αυτή που ζητήσαμε από τις νομικές υπηρεσίες που θέλησαμε να συμβουλευτούμε. Και είναι σαφές επίσης ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μετά την ψηφοφορία στην νομική επιτροπή που είναι καθήλυνα αρμόδια. Οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε προηγουμένως. Πρότεινα λοιπόν, αν δεν ψηφίσουμε σήμερα, να ψηφίσουμε κάποια στιγμή στο Στρασβούργο. Δηλαδή τρει-τέσσερι μέρε πριν την νομική επιτροπή για να μπορέσουμε να στείλουμε την γνωμοδότησή μα. Με τα λόγου γνώσεω. Να μας έχει δώσει την άποψή της λοιπόν νομική υπηρεσία και να προλάβουμε και το θέμα της νομικής επιτροπής. Ευχαριστώ. Πράγματι έφτασε ένα μήνυμα από τη γραμματεία της κυρίας Ρέγνερ όπου λέγεται ότι θα πρέπει να ψηφιστεί σήμερα η γνωμοδότηση. Αν πράγματι πρέπει να κάνουμε δεκτή την πρόταση αυτή, αυτό δεν θα γίνει την Τετάρτη, Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα για να μην μπερδευόμαστε, ας περιμένουμε την κυρία Ρέγνερ να μας εξηγήσει τι θα κάνουμε τελικά. Περνάμε στο ένατο θέμα, τροποποίηση του άρθρου 70 του κανονισμού για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια των νομοθετικών διαδικασιών. Έχει ζητηθεί να επανεξεταστούν οι κανόνες οι σχετικοί με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης. Έγινε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ζητήθηκε από τον συνάδελφο Γκουερέρο να κάνει την έκθεση και θα πρέπει ο εισηγητής σήμερα να μας παρουσιάσει σε μια πρώτη φάση την έκθεσή του. Έχει συναντηθεί και με ε, τους εκπροσώπους της διάσκεψης των Προέδρων και με κάποια μεμονωμένα μέλη. Γκουερέρο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξετάζουμε την ανάλυση μιας πιθανής αναθεώρησης του άρθρου 70 όσον αφορά τις συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση. Η πρώτη φορά που το κάναμε ήταν με ένα έγγραφο εργασίας που εγώ είχα υποβάλει στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο εργασίας ευρέως τροποποιήθηκε και καθώς ε, μεταμορφώθηκε στην προσωρινή έκθεση, draft report, σχέδιο έκθεσης, υπέστη σημαντικές αλλαγές με τρόπο που θα συμβούλευα να ξεχάσουμε αυτό το έγγραφο εργασίας κατά κάποιο τρόπο και να δούμε μόνο αυτό που αναφέρεται στο σχέδιο ε, έκθεσης. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω κάτι άλλο. Είχα επαφές και συνεδριάσεις πράγματι ουσιαστικά με κάποιους από τα μέλη των ξεχωριστών ομάδων για αυτό το θέμα και παρουσιάστηκα επίσης και στην διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και υπέβαλα τις ουσιαστικές γραμμές αυτής της έκθεσης που παρουσίασα. Είχαμε την Προεδρία επίσης και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, της δικής μας Επιτροπής, μια συνάντηση με ηγέτες επικεφαλής ομάδων στο σώμα στην Ευρωβουλή. Επίσης συνήλθα με κάποιους εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές, όπως την κυρία Γιαννάκου παράδειγμα. Και στο τέλος τέλος εκπώνησα αυτή την προσωρινή έκθεση. Πρέπει επίσης να επισημάνω και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσω αυτό, ότι αυτή δεν είναι μια έκθεση για το αν είναι καλό ή όχι, αν είναι σκόπιμο ή όχι να ξεκινήσουμε προσεγγίσεις σε ε, διαδικασίες πρώτης ανάγνωσης. Είναι ένας προβληματισμός ή μια απόφαση που ξεπερνά τα όρια αυτής της έκθεσης. Αυτή η έκθεση είναι μόνο στην περίπτωση εκείνη όπου ληφθεί, ληφθεί απόφαση να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης σε πρώτη ανάγνωση τότε να δούμε υπό ποιου όρου και προποθέσει που πρέπει να εντάξουμε και να δούμε από τον κανονισμό για να διασφαλίσουμε ότι πέρα από την αποτελεσματικότητα τη διαπραγματευτική θα είναι σεβαστή και η διαφάνεια. Θα είναι σεβαστή και η πληροφόρηση και η ενημέρωση των διαφορετικών ομάδων και θα είναι σεβαστή η δυνατότητα να παρεμβαίνει κανείς κατά τη διάρκεια όλης συνολικά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Το επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό γιατί σε κάποιες αποσυζητήσεις που είχα Είδαμε ότι ξεκινά διαβούλευση και συζήτηση αν θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση στην πρώτη ανάγνωση ή στη δεύτερη ανάγνωση ή στη συνδιαλλαγή. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό το θέμα λοιπόν αναφέρεται στο πώς θα διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και θα υπάρχει λογοδότηση σε σχέση με διαπραγματεύσεις στη διαδικασία πρώτης ανάγνωσης. Όπω γνωρίζετε, Πρόεδρε, εσεί και όπω γνωρίζουν και τα μέλη αυτή τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ο λόγο για τον οποίο προσεγγίζουμε αυτή την αναθεώρηση του κανονισμού είναι ακριβώ επειδή η διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών σε μια προηγούμενη στιγμή και υστερότερα μετά από αυτήν η διάσκεψη των Προέδρων Ομάδων <clears throat> κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αρκετά συχνά στις διαδικασίες ε, διαβουλεύσεων και διαπραγμάτευσης το υπόλοιπο των ομάδων που, στις οποίες δεν ανήκε ο διαπραγματευτής είχαν πολύ αραιές ε, ή καθόλου πληροφορίες για τη διαπραγμάτευση και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και οι πολιτικές ομάδες στο σύνολό τους έπαιρναν αυτές τις πληροφορίες μόνο ή μπορούσαν να πάρουν αυτές τις πληροφορίες όταν ερχόταν η στιγμή ψήφισης στην Ολομέλεια μόνο. Έτσι λοιπόν, ας το πούμε έτσι, υπήρχε μια θολή διαδικασία όσον αφορά την διαπραγμάτευση για όσους δεν ε, εμπλεκόντουσαν σε αυτήν. Και έτσι δεν μπορούσαν οι ομάδες να αντιδράσουν έγκαιρα. Σαν αποτέλεσμα προβληματισμών και σκέψεων όσον αφορά την διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών και ε, από πλευρά του, ο πρόεδρο του, ο του Κοινοβουλίου απέστειλε στον πρόεδρο τη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπής ένα αίτημα Έτοιμα για την ανάγκη ή τη σκοπιμότητα να μεταθέσουμε, μεταφέρουμε από τον δεοντολογικό κώδικα κάποιες από τις αρχές ε, του κανονισμού, ώστε να γίνουν υποχρεωτικού χαρακτήρα κάποια πράγματα, εντάσσοντας, εντάσσοντας αυτά στον κανονισμό όσον αφορά προβλέπει προϋποθέσεις και όρους που αυτή τη στιγμή δεν έχει υποχρεωτικού χαρακτήρα τέτοιες διατάξεις ο δεοντολογικός κώδικας, ώστε να συμπληρωθεί έτσι. Με αυτόν τον τρόπο εγώ εκπώνησα τελικά αυτή την έκθεση και έχουμε δύο κατηγορίες ζητημάτων εδώ που είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους αυτές οι δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά την ένταξη στον κανονισμό αυτών των αρχών της, ε, του κώδικα δεοντολογίας για την οποία αυτή η κατηγορία δεν φαίνεται να υπάρχει σύμφωνα με τις συζητήσεις που είχαμε εδώ για το έγγραφο εργασίας δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα από πλευρά των μελών της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και έχουμε ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι πιο, ε, περισσότερο υποσυζήτηση και προβληματικό. Ποιος θα είναι ο ρόλος στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και ποιος θα είναι ο λόγος που θα έχουν επιμέρους ατομικά οι ευρωβουλευτές, οι ενωμένοι σε ομάδες ευρωβουλευτές όσον αφορά την εντολή για διαπραγμάτευση. Με τέτοιο τρόπο ώστε <clears throat> αν μέλη της Επιτροπής, για παράδειγμα, έχουν διαβάσει αυτή την έκθεση, την, το σχέδιο έκθεση, την προσωρινή έκθεση που έχω υποβάλει, θα δουν ουσιαστικά το εξή περιεχόμενο, το εξής συμπέρασμα. Πρώτα απ' όλα, λέμε ότι η απόφαση του να ανοίξουν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σε πρώτη ανάγνωση μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιτροπή, όποια και αν είναι αυτή. Αυτή η απόφαση θα πρέπει να εμπεριέχει υποχρεωτικά μια εντολή διαπραγμάτευση. Είτε με κάποιες τροπολογίες, τοποποίησει, ή με τον καθορισμό κάποια σειρά προτεραιοτήτων ή κάποιων προσανατολισμών Αφετέρου, όπως θα μπορέσετε να δείτε, πρόκειται για μια ευέλικτη διαδικασία. Σε κάποιες δηλαδή περιπτώσεις αυτή η εντολή θα μπορεί να εμπεριέχει σαφώς και αλλαγές, τροποποιήσεις <clears throat> σε άλλες, άλλες φορές ε, προσανατολισμούς ή αρχές όσον αφορά την ε, διαπραγμάτευση. Αυτή επίσης η απόφαση θα πρέπει να έχει, να εμπεριέχει και το θέμα της ομάδας διαπραγμάτευσης ομάδας διαπραγμάτευσης. Εδώ τι καθορίζουμε. Προσδιορίζεται ότι ως αρχή οι διαπραγματεύσεις αυτές ως θέμα θα πρέπει να, στοχεύ, να βρίσκονται υπό την εντολή, υπό την ε, ε, πρωτοκαθεδρία του Προέδρου της Αρμόδιας Καθήλην Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχε τεθεί στους Προέδρους ε, των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Εκεί είχε πρωτοπαρουσιαστεί, βρήκε πολύ μεγάλη ευρύτατη υποστήριξη εκεί και έχει και ένα τελικό στόχο πολιτικά. Δηλαδή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκπροσωπεί το σύνολο μιας, των μελών μιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και έτσι μπορεί να δώσει εντολή στον εισηγητή ή μπορεί να δώσει εντολή σε έναν αντιπρόεδρο της Συνοβουλευτικής Επιτροπής να έχει την αρμοδιότητα και πρωτοκαθεδρία σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όμως, καταρχήν ως θέμα αρχής, η πολιτική ευθύνη για αυτές τις διαπραγματεύσεις θα είναι θέμα που θα υπομίζεται ο ίδιος ο πρόεδρος αυτής της αρμόδιας καθήλυν, δηλαδή Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Εκείνος θα μπορεί να δει αν θα πρέπει και αν θα θέλει να δώσει αυτή την εντολή σε κάποια άλλα μέλη της Κοινοβουλευτικής του Επιτροπής ή στον εισηγητή σε κάποιον από του αντιπροεδρού ώστε αυτό να διαπραγματευτεί ώστε με τέτοιο τρόπο και η εντολή και το περιεχόμενο της εντολής από τη μια πλευρά, όπως από την άλλη πλευρά και η σύνθεση της Επιτροπής που θα διαπραγματεύεται, πρέπει επίσημα να έχει καθοριστεί με απόφαση της αρμόδιας καθήλυν Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Προτού δηλαδή προχωρήσουμε ή ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία διαπραγμάτευσης σε πρώτη ανάγνωση. Πρέπει αυτά να έχουν διασφαλιστεί. Αυτές αυτή η απόφαση της Επιτροπής λοιπόν μεταφράζεται και θα μεταφράζεται στις διάφορες γλώσσες. Θα διαβιβάζεται στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε όλους τους ευρωβουλευτές. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου στην αρχή, κατά την έναρξη των εργασιών της επόμενης Ολομέλειας μετά από την ε, λήψη αυτής της επιστολής γνωστοποίησης θα το γνωστοποιεί αυτό στα μέλη, στους ευρωβουλευτές. Και αν από τα μέλη τους ευρωβουλευτές δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση ή ένσταση, θα θεωρείτε ότι επικυρώνεται, ότι εγκρίνεται η εντολή προς διαπραγμάτευση. Και έτσι θα θεωρειται οτι θα εγκρίνεται η έναρξη αυτών των διαδικασιών. Δεν θα... Ε, αυτό το θέμα είναι ένα σημαντικό θέμα και δεν θέλω να το αναμειγνύουμε με το θέμα επί του οποίου υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση. Λοιπόν, έχοντας καθορίσει ότι η εντολή για διαπραγμάτευση θα έχει με αυτόν τον τρόπο αποσαφινιστεί και η ομάδα που θα διαπραγματευτεί θα έχει καθοριστεί, θα ενημερώνει αυτή η ομάδα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή μετά από κάθε ε, τριμερή διάλογο. Τα κείμενα τα οποία θα είναι υποσυζήτηση θα γνωστοποιούνται και θα γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα στα μέλη της Επιτροπής. Αν υπάρχουν κάποιοι λόγοι ε, ε, ιδιαίτερα επίγοντος χαρακτήρα, θα γνωστοποιούνται αυτά τα θέματα στην Προεδρία, στους κοιόδης εισηγητές και στους συντονιστές, στους και στους συντονιστές των διαφορετικών ομάδων. Ο γενικός ε, κανόνας είναι ότι μετά από κάθε τριμερή διάλογο θα ενημερώνονται όλα τα μέλη της Επιτροπής. Η εξαίρεση θα είναι για επίγοντες λόγους να μπορούν να, σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις να ενημερώνονται ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οι σκιώδεις συζητητές και οι συντονιστές. Εφόσον θα έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο κάποια στιγμή και πάλι οι συντονιστές θα ενημερώνονται άμεσα και το σύνολο των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα εξετάζει την ε, συμφωνία που θα είχε επιτευχθεί και θα υποβάλλεται στην Ολομέλεια ως έκθεση υπομορφή, ας το πούμε, έκθεσης ε, σε σχέση κιόλας και με προτάσεις ε, τροποποίησης που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο συγκεκριμένο κείμενο. Για λόγους επίγοντος χαρακτήρα, αν αυτό δεν είναι δυνατό να γίνεται, θα υποβάλλεται στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στον εισηγητή, στους κοιόδης εισηγητές και στους συντονιστές. Υπάρχει και ένα ίσονο σημασία θέμα για τι συναρμόδιε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Όταν υπάρχουν τέτοιε συναρμόδιε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού και σε ίσε κοινέ συνεδριάσει, σύμφωνα με το 51, το άρθρο 51, και οι δύο ή οι περισσότερε επιτροπέ πρέπει να είναι και εκείνε σύμφωνε για την έναρξη διαπραγματεύσεων και την εξέλιξή του και στην περίπτωση που δεν θα συμφωνούν, η Προεδρία της Διάσκεψης των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα λαμβάνει σχετικά απόφαση για τον πρακτέ, περί των πρακτέων. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα της Ολομέλειας. Αν θα το θυμόσαστε ίσως, το θέμα που είχε τεθεί ήταν, αν δεν υπήρχε, αν δεν υπάρχει καμιά αντίδραση όσον αφορά τις πληροφορίες, την ενημέρωση που υποβάλλεται, που δίνεται από τον πρόεδρο της ε, ε, του Κοινοβουλίου στην έναρξη των εργασιών, η ομάδα για τη διαπραγμάτευση αυτή και η εντολή θα θεωρούνται ότι έχουν επικυρωθεί. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων μπορεί να υπάρξει μια αντίδραση, ώστε να συζητηθεί στην Ολομέλεια και ενδεχόμενα να υπάρξει κάποια αναθεώρηση ή τροποποίηση της εντολής ή της σύνθεσης της διαπραγματευτικής ομάδας. Στην δική μου έκθεση <clears throat> η δυνατότητα του να εξεταστεί αυτό το θέμα Ω εντολή, ω αρμοδιότητα δίνεται στη διάσκεψη των προέδρων, διάσκεψη των προέδρων ομάδων, των κοινοβουλευτικών ομάδων, που μπορεί να εξετάσει το θέμα μια ψήφισή στην Ολομέλεια για επικύρωση ή τροποποίηση της εντολή διαπραγματευτικής εντολή. Εγώ στι επαφέ και συζητήσει που είχα, έχω συνειδητοποιήσει βέβαια ότι υπάρχει κάποια θέση η οποία λέει ότι θα επιθυμούσαν, θα ήταν ευκταίο, όχι μόνο η διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών να μπορεί να θέτει στην Ολομέλεια αυτό το θέμα, αλλά επίσης να μπορεί να γίνεται αυτό, ας το πω έτσι, και από κάποιες ομάδες ή από ένα σύνολο αριθμού ευρωβουλευτών που θα έχουν συναθριστεί πέρα αυτού. Εγώ σε σχέση με αυτή την δυνατότητα θα ήθελα να πω ότι το μόνο σκεπτικό, η μόνη σκέψη που θα έπρεπε να μας εμπνέει σε αυτό το θέμα είναι ότι σε όλες τις συνεδριάσεις στις οποίες εγώ μπόρεσα να συμμετάσχω και παρακολούθησα, σε όλες εκείνες που αντάλλαξα απόψεις με άλλους για αυτό το θέμα, υπήρχε σύμπτωση απόψεων για το ότι δεν θα έπρεπε να διευκολύνουμε όλες οι διαπραγματευτικές εντολές να μπορούν να τίθενται υπό και επανεξέταση στην Ολομέλεια, να αναθεωρούνται στην Ολομέλεια, να επαναπέμπονται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να ξεκινά μια διαδικασία δούνε και λαβίνω όπου θα υπάρχει ανταλλαγή διαρκώς απόψεων που θα υπονομεύει και την ίδια την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου που όταν έρχεται η στιγμή να λαμβάνονται αποφάσεις και μάλιστα κατεπηγόντως να αρχίζει να παίζει το μπαλάκι να περνάει από την Ολομέλεια προς την Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν ε, έχω πρόθεση να ε, αναφερθεί για το ότι ποιε θα έπρεπε να είναι οι προποθέσει, ε, οι απαιτήσει, ο αριθμό βουλευτών κτλ. Αλλά θα έπρεπε να πω ότι δεν πρέπει να είναι μια πρόταση που αν θέλει κάποια ομάδα να το κάνει αυτό θα διευκολύνει απόλυτα το να αναθεωρούνται οι εντολές ανά η στιγμή εντολές για διαπραγμάτευση προς κάποια κοινοβουλευτική επιτροπή. Τούτων λεχθέντων ολοκληρώνω και λέγω υπάρχει ευρεία συνένεση για αυτά τα οποία αναφέρονται στην επίσημη και τυπική έγκριση όσον αφορά την διαπραγματευτική εντολή και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής επιτροπής που θα κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις και που πολιτικά θα είναι αρμοδιότητα της του Προέδρου αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα μπορεί να τη μεταθέτει στον Αντιπρόεδρο, στον εισηγητή κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία επ' αυτών των θεμάτων. Μετά από κάθε συνάντηση, κάθε τριμερή διάλογο θα υπάρχει ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και όταν θα υπάρχει συμφωνία θα πρέπει επίσημα να επικυρώνεται, να εγκρίνεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή προτού διαβιβάζεται στην Ολομέλεια για ε, ψήφιση και τελική έγκριση. Πιστεύω, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποια δυνατότητα κάποια ευελιξία όσον αφορά τους όρους και τις προποθέσει υπό τις οποίες και τους οποίους μπορεί να ε, ζητηθεί να αναθεωρείται αυτή η εντολή στην ε, Ολομέλεια. Και όπως επεσήμανα τελικά στο τέλος τέλος προσβλέπω και αναμένω να δω ποιες θα είναι οι τροπολογίες από πλευρά των ομάδων για αυτό το θέμα. Και συνιστώ θα θέλω να συστήσω υπό το δικό μου πρίσμα μια τέτοια τροπολογία να μπορεί να, μια τέτοια τροποποίηση να διασφαλίζει το ότι δεν θα είμαστε παρατηρητές μιας διαρκούς ε, διαδικασίας ε, ε, από δυνάμωσης και ίσως και υπονόμευσης αυτών των διαδικασιών και εντολών σε σχέση με την Ολομέλεια. Γνωρίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο παρουσίασα τις αδρές γραμμές, ουσιαστικές γραμμές αυτής της έκθεσης και σε σχέση με την πλειοψηφία των προέδρων της, ε, των κοινοβουλευτικών επιτροπών, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε χωρίς να απομένουν θέματα που εκκρεμούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ε, συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντική έκθεση και πολλές οι για, και, την τροποποίηση του κανονισμού στο άρθρο 70. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν αφορά μόνο ε, τη συμφωνία σε πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση, αλλά όλες τις νομοθετικές διαδικασίες και ιδιαίτερα τη διαδικασία της συναπόφασης. Επιπλέον, η δευτερη αναγνωση αλλα ολες τι νομοθετικες διαδικασιες και ιδιαιτερα τη διαδικασια της συναποφασης επιπλεον κανόνες που διέπουν τις διοργανικές ε, συνεργασίες μπορεί να είναι επίμαχες, το, ε, ε, επίμαχοι κανόνες και οι διαδικασίες. Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα να ξεπεράσουμε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και μονοσήμαντο κυρίως προς το Συμβούλιο. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις επί του προτινομένου κειμένου. Πρώτον, υποστηρίζω την ιδέα ότι θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός και οι κανόνες και να γίνει ε, νομικά δεσμευτικό. Ε, να λαμβάνεται υπόψη ο, ο κώδικας διοντολογίας και μπορούμε να ε, το ορίσουμε αυτό ρητά όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να βρίσκει εφαρμογή ο κώδικας διοντολογία. Το είπε και ο εισηγητή ε, ξεκάθαρα. Για την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να υπάρχει μια απόφαση ε, αρκετά σαφής και να ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει. Να είναι και η εντολή αλλά και η σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Όσο και το πεδίο εφαρμογής. Αυτό λίγο με ανησυχεί. Έτσι, το πεδίο εφαρμογής της εντολής. Ποια θα είναι αυτή η εντολή. Θα πρέπει να είναι πολύ καλά περιγεγραμμένη και να λαμβάνει ε, ε, λέτε διαφορετικές μορφές. Αυτό δεν μου αρκεί ως διατύπωση. Ή αυτές οι μορφές θα πρέπει να ε, κατονομάζονται ρητά ή να μην αναφέρονται καθόλου. Αλλιώς, αντί να διευκρινίσουμε το κείμενο και να το κάνουμε πιο σαφές, θα το θολώσουμε ακόμα περισσότερο. και θεωρώ σωστό ε, δίκαιο να είναι επικεφαλής ε, της διαπραγματευτικής ομάδας ο πρόεδρος της Επιτροπής ή κάποιος αντικαταστάτης που θα τον έχει ορίσει ο ίδιος. Ωραία όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να ε, πούμε και τα μέλη ποια θα είναι. Ο ίδιος ο κώδικας δεν είναι αρκετά σαφής για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. επίση και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί και να αναφέρεται ρητός μοναδική απόφαση ε, της Επιτροπής για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Και θα πρέπει, λέτε, να διαβιβάζετε στον Πρόεδρο και να διανέμετε σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό είναι σαφές ότι χρειάζεται μετάφραση. Δεν υπάρχει ανάγκη να ε, γραφτεί ρητά ότι χρειάζεται μετάφραση. Γι' αυτό ε, προτείνω να απαλληφθεί αυτό το τμήμα της συγκεκριμένη τροπολογίας. Επιτρέψτε μου τώρα να πω δύο λόγια για τρει-τέσσερι τροπολογίες. Η τροπολογία υπερθούν τρία. Φοβούμαι ότι δεν μπορώ να καταλάβω αρκετά την πρότασή σας για τη δράση που μπορεί να αναλάβει το Κοινοβούλιο αφού θα έχει ε, λάβει την απόφαση της Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής τι αφορά την εντολή και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Έτσι δεν είναι. Όταν λαμβάνει την απόφαση η Επιτροπή μπορεί να τη λαμβάνει μόνο ως σύνολο. Εκτός αν έχει αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων, ε, οπότε και θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε από το γεγονός αν θα πρέπει να αρχίσουν καν οι διαπραγματεύσεις. Αν αποφασίσει μια επιτροπή, ας πούμε, και κληθεί να ψηφίσει και η Ολομέλεια και την απορρίπτει, τι σημαίνει αυτό. Δεν θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Μα είναι το ίδιο πράγμα. Χρειάζομαι περισσότερες εξηγήσεις. Αν αυτό είναι σύγκρουση ή όχι αρμοδιότητα. Έρχομαι τώρα στην τροπολογία 4. Είναι σαφές γενικό ότι η ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια πρέπει να είναι δεδομένη. Γι' αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται από τη διαπραγματευτική ομάδα η Επιτροπή. και στον πρόεδρο, στους σκιώδεις ηγητές και τους συντονιστές αν θέλετε, όχι σε όλη την Επιτροπή. Έχω όμως σοβαρές αμφιβολίες και φοβούμε ότι αυτή η εξέλιξη θα γίνει κανόνας. Να μην την επιτρέψουμε. Αλλιώς δεχόμαστε παραβίαση του κανονισμού. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε ακριβώς τι εννοείτε. Ε, να είναι τακτική ενημέρωση. Κάθε πότε δηλαδή θα γίνεται. Ε, ο στόχος είναι και η διαφάνεια και ε, στην τροπολογία όμως 5 λέτε να ενημερώνονται μόνο οι ε, συντονιστές εάν οδηγούμαστε σε συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Γιατί μόνο οι συντονιστές. Αν μη τι άλλο και οι σκιώδεις συγητές θα πρέπει να ενημερώνονται. Γιατί οι σκιώδεις συγητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες και ε, οφείλουν να είναι ενήμεροι κατά την άποψή μου. Τροπολογία 6. Η διαδικασία υποβολή σχεδίου νομοθετικής πράξης από την Επιτροπή είναι και αυτή συγκεχημένη και μπερδεμένη. Δεν έχω καταλάβει ποιος εγκρίνει το συμβιβασμό, το σύνολο της Επιτροπής. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν πιστεύετε ότι είναι περίπλοκη αυτή η μορφή εκπροσώπησης. Και να υποβάλλεται ο συμβιβασμός προς εξέταση στην Ολομέλεια. Αν πάλι θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται ολόκληρη επιτροπή, αλλά ένα τμήμα της επιτροπής, ποιο θα είναι αυτό. Και θα πρέπει να το έχει εγκρίνει αυτό το τμήμα, το υποσύνολο. Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό, αλλά δεν είναι διαφανές. Επίσης, υπάρχει και μια σαφής διαδικασία για το διακανονισμό των ε, διαφορών ε, περί αρμοδιοτήτων και θα πρέπει να ξαναδούμε την τροπολογία 6. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε αλλαγές μόνο στο άρθρο 70. Τι εννοώ συγκεκριμένα. Σε περίπτωση διαφωνίας για το εάν θα πρέπει να ξεκινήσουν και να διεξαχθούν ε, διαδικασίες. Αυτό δεν θα πρέπει να το αποφασίζουν οι πρόεδροι των επιτροπών, αλλά και οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων, σύμφωνα με το άρθρο 188, εδάφιο 2. Τελική παρατήρηση. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι για τη συνολική διαδικασία. Ε, τα άρθρα 50 και 51 του κανονισμού και καμιά φορά και το 49 μπορεί να βρίσκουν εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή αυτή θα πρέπει να διευκρινίζεται γενικώ. Και όχι να, να εξηγούμε πώς εφαρμόζονται το άρθρο 50, αλλά λέμε μουτά μουτάτης μουτάντης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτά ήταν τα σύντομα σχόλιά μου. Ο κύριος Ντάφ έχει ζητήσει το λόγο. Very good. Um, I'd also like to και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκουερέρο για την εξαιρετική του δουλειά. και συμφωνώ με την πρόθεσή του να προστατεύσει τα, θα έλεγα, τα συμφέροντα καλώς εννοούμενα των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να καταστήσει ακόμα περισσότερο υπεύθυνο τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών που συμμετέχουν και παρακολουθούν γενικότερα την νομοθετική προσπάθεια την οποία κάνει το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση βασικά για την πρώτη τροπολογία. βάζετε μια ρήτρα στο τέλος, λέγοντας ότι το άρθρο αυτό δεν θα ισχύσει για τις ανεπίσημες επαφές ε, πρώτου επίπεδου ή διερευνητικές με το Συμβούλιο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το, ε, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον. Δεν θα πρέπει δηλαδή να αυτοπεριοριστούμε εν πολλής σχετικά με κάποιες ε, ε, συζητήσεις και με κάποιες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο οι οποίες δεν είναι επίσημες. Πρέπει να μην περιοριστούμε θα έλεγα. Αν συμπεριλάβουμε μια τέτοια ρήτρα όπως αυτή την οποία προτείνεται στην ουσία δημιουργείται κάποια προβλήματα και τίθενται ερωτηματικά για το εύρος και την σημασία αυτού του είδους των διερευνητικών επαφών. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η σιωπή είναι η καλύτερη λύση. Mm. Ευχαριστώ κύριε Ντάφ. Η κυρία Γιαννάκου, αλλά θυμίζω ότι η κυρία Γιαννάκου να έχει ζητήσει το λόγο. Θυμίζω ότι στις 10 θα ξεκινήσουμε ε, ψηφοφορία. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα σας ακούσουμε λοιπόν, αλλά σύντομα, κυρία Γιαννάκου. Πρόεδρε, το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί θέλουμε να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε το άρθρο 70 του κανονισμού διότι αν δεν καθοριστεί ο στόχος, φυσικά ο καθένας μπορεί να θέλει να αλλάξει ό,τι θέλει. Παρατηρείται το φαινόμενο πρώτον, οι βουλευτές λόγω του μεγέθους του Κοινοβουλίου να μην μπορούν να παρακολουθήσουν καθόλου και ιδιαίτερα οι μικρές εθνικές ομάδες να μην μπορούν καθόλου να παρακολουθήσουν τι γίνεται στο Κοινοβούλιο. Δεύτερον, πολλά μέλη των επιτροπών δεν μπορούν να παρακολουθήσουν καν τι γίνεται στις επιτροπές δημιουργούνται ομάδες εργασίας, αποφασίζουν μόνοι τους οι πρόεδροι, οι συντονιστές κτλ. Αυτό τι σημαίνει. Ότι το κοινοβούλιο δεν συμμετέχει. Απόδειξη αυτού είναι το φαινόμενο του κοινοβούλιο να έχει γίνει ένα είδος θεάτρου όπου σε όλους τους διαδρόμους του γίνονται διάφορες απίθανες εκδηλώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική ή με την Ευρώπη γιατί θέλουν να εκφραστούν με κάποιο τρόπο ή θέλουν να εκφραστούν προς τις εθνικές τους αρχές. Αν θέλουμε να μας πάρουν στα σοβαρά καταρχήν τα άλλα όργανα, θα πρέπει πρώτον να έχει ρόλο η Ολομέλεια. Εάν δεν έχει ρόλο η Ολομέλεια, δεν υπάρχει πολιτικό βάρος. Δεύτερον, να έχει ρόλο η Επιτροπή, επομένως τα μέλη της Επιτροπής να, να γνωρίζουν πλήρως, μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες. Σε όλες τις γλώσσες, κύριε Πρόεδρε το κείμενο που αποφασίζεται καθώς και εντολή που δίνεται στη διαπραγματευτική ομάδα. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να μας πάρουν στα σοβαρά. Τρίτον, οι επιτροπές κάποτε πρέπει να αποφασίσουν να αναπέμπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που έρχονται για συνεχείς αλλαγές επικειμένων νομοθετικού περιεχομένου που έχουν αλλαγεί την προηγούμενη χρονιά παραδείγματος χάρη δεν είναι δυνατόν εδώ να δημιουργείται, να διευρύνεται τεχνητά ο κύκλος εργασιών και ό,τι στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ να εγκρίνεται. Κάποτε πρέπει να πάρουμε το θάρρος να επιστρέψουμε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί σοβαρά, δεν έχουν εξεταστεί σε βάθος και προσβάλλουν το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό δεν γίνεται πουθενά. Η προσπάθεια του κυρίου Γκερέρο είναι πολύ σοβαρή. Δεν καλύπτει όμως το θέμα της Ολομέλειας κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να αποφασίζει τα πάντα. Αλλιώ το Κοινοβούλιο καταργείται. Και η κοινοβουλευτική τάξη και η δημοκρατία καταργείται. Μόνο η Ολομέλεια μπορεί να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί κάτι ή εάν θα το αναπέμψει σε επόμενη σύνοδο προκειμένου να υπάρξουν τροπολογίες από την Ολομέλεια έτσι λοιπόν η πρόταση να υπάρχει ένας αριθμός βουλευτών ή πολιτικών ομάδων, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί μπορεί μικρές πολιτικές ομάδες κατά κάποιο τρόπο να προσπαθήσουν να εμποδίσουν το έργο του Κοινοβουλίου. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει κάποιος τρόπος με κάποιο εύλογο αριθμό βουλευτών ή πολιτικών ομάδων που να μπορούν να κάνουν αποδεκτό ή όχι να αρνηθούν την αποδοχή και να αναπέμψουν σε επόμενη ολομέλεια το κοινοβούλιο δεν έχει κύρος και βεβαίως εγώ προσωπικά δεν συζητώ αυτό που γράφεται ότι αν η Επιτροπή δεν προλάβει θα αποφασίζουν οι συντονιστές και ο πρόεδρος της Επιτροπής και θα ενημερώνονται και θα έχετε στην Ολομέλεια. Αυτό κύριε πρόεδρε προσβάλλει τελείως την κοινοβουλευτική τάξη. Δηλαδή ποιος θα φέρει στην Ολομέλεια ένα θέμα. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Σε κανένα κοινοβούλιο του κόσμου δεν θα το βρείτε αυτό και ομολογώ ότι αυτό το συγκεκριμένο άρθρο εμένα προσωπικά με σοκάρει. Ότι δηλαδή είναι δυνατόν αδιαφανώς χωρίς να γνωρίζει η Επιτροπή να έρθει κάτι στην Ολομέλεια. Τότε περνάμε σε μια διαδικασία όπου κανείς δεν γνωρίζει ποιος αποφασίζει τι και τι κάνει και ποιος αποφασίζει στο τέλος. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο φυσικά. Διότι κανείς δεν θα πάρει στα σοβαρά ένα κοινοβούλιο το οποίο θεωρεί πιο σημαντική τη βιασύνη για να δοθεί μια απάντηση από την ουσία του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γιαννάκου. Ο Μέντες Βίγκο έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η περίπτωση που μας απασχολεί είναι Μία ε, περίπτωση μετάλλαξης ε, τη χαρακτηρίζω, όπως λένε τα εγχειρίδια. Μετά τη συνθήκη του Μαστρίχτ είχαμε τρεις αναγνώσεις, μετά φτάσαμε σε δύο αναγνώσεις συν συνδιαλλαγή και έχει έρθει η στιγμή που διαπιστώνουμε ότι αυξάνονται τα ποσοστά των νομοθετημάτων που περνούν από το Κοινοβούλιο και λύνονται σε πρώτη ανάγνωση. Γιατί, για τους εξής δύο λόγους πιστεύω εδώ. Πρώτον, γιατί υπάρχει ανάγκη να δρούμε ε, γρήγορα και αποτελεσματικά και δεύτερον, διότι και δομικά, διαρθρωτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρωθούν τα κριτήρια που ορίζει η συνθήκη για να εγκριθούν με απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση τροπολογίες. Λοιπόν, προσπαθούμε να πατρέψουμε τώρα την πολιτική και την αποτελεσματικότητα και γι' αυτό καταλήγουμε, καταφεύγουμε σε ε, συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση. Και ακριβώς επειδή τώρα έχουμε μια μεταβατική κατάσταση ε, που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό, χρειάζεται τροποποίηση και μάλιστα με μεγάλη αφοσίωση και μεγάλο ταλέντο ο κύριος Γκερέρο μας προτείνει ε, μια λύση με τις άλλες πολιτικές ομάδες για να μην περιπλέξουμε υπερβολικά τα πράγματα και να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στη λήψη των αποφάσεών μας. Ωραία. Συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε. Ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι ε, πιέζει ο χρόνος, αλλά δεν θα επαναλάβω τα σημεία στα οποία συμφωνώ, που είναι σχεδόν όλα. Ε, ο κώδικα συμπεριφορά και δεντρολογία να ενταχθεί στον κανονισμό μου φαίνεται σωστό αυτό. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι ίσω πιο επίμαχο είναι το θέμα τη εντολή. Επ' αυτού, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορα πράγματα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία για το κείμενο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή που είναι αρμόδια. Η εντολή είναι το κείμενο της Επιτροπής. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Που θα το στείλουμε στην Ολομέλεια. Μια συμφωνία μιας Επιτροπής δεν θα είχε νόημα. Στην πραγματικότητα τι συζητούμε. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή δεν αποφαίνεται ακόμα και οι διαπραγματευτές έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το Συμβούλιο. Ε, το έχουμε ζήσει αυτό στην νομοθετική πρωτοβουλία των πολιτών στην πρωτοβουλία των πολιτών και ψηφίσαμε μια γενική εντολή στην Επιτροπή. Ε, με ποιον άλλο τρόπο, γενική θα είναι η εντολή. Εμπιστευόμαστε τους εισηγητέ και τους λέμε αυτοί είναι οι ε, προσανατολισμοί, οι κατευθυντήρες γραμμές και πηγαίνετε. Γιατί πάντα στο τέλος αυτή εδώ η Επιτροπή και η ολομέλοι ενδεχομένω έχουν την πολιτική δυνατότητα να απορρίψουν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Ε, ας μην υπερβάλλουμε τώρα και στη σημασία της εντολής. Κυρία Γιαννάκο, ε, την πολιτική απόφαση τελική την έχει πάντα η Ολομέλεια, γιατί μπορεί να απορρίψει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο θα διαμορφώσουμε αυτή την εντολή για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη συμμετοχή, να γνωρίζουμε όλοι τι διαπραγματεύονται οι διαπραγματευτές μας. Στην Οικονομική Επιτροπή έχω συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις και ο πρόεδρος της Επιτροπής, οι συντονιστές, οι σκιώδεις. Ήταν το σχήμα και λειτουργήσε αρκετά καλά. Πάντα αισθανόμουν πολύ άνετα, ενταγμένο στο σχήμα και οι εξηγήσει ήταν ε, πάρα πολύ ικανοποιητικέ. Τελικά, τι θέλουμε. Να συμμετέχουν τα μέλη της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορώ ε, φίλε Γκαργάνη, δεν, μπορώ να συνεχίσω να μιλάω. Ράνι. Το άρθρο 70 βλέπετε παθιάζει τον κόσμο. Άμα μιλάω στο τηλέφωνο δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, τι έλεγα κύριε Πρόεδρε, έχω χάσει τον ερμό μου τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ε, τι έλεγα Πρόεδρε. Θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να συμμετέχουν, λέτε, τα μέλη της Επιτροπής, οι βουλευτές. Επιμένω, όταν δεν έχει υπάρξει ακόμα ψηφοφορία και απόφαση της αρμόδιας επιτροπής και έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις. Αν υπάρχει πλειοψηφία να πάει στην Ολομέλεια, θα πρέπει να δούμε πώς θα έχει διαδικασία αλλά και ποιοι θα δικαιούνται να ζητήσουν επανάληψη και επανεξέταση να το σκεφτούμε αυτό. Γιατί μπορεί να σημαίνει ένα καθεστώς συνέλευση. Ας πούμε, εγκρίνει η Επιτροπή μια εντολή ε, πριν να έχει αποκριστηλωθεί αυτή σε τροπολογίες και στο κείμενο. Και πάμε στην Ολομέλεια. Πρώτον, ποιο μπορεί να επανεξετάσει, ποιο μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση, πόσε πολιτικέ ομάδε ή πόσοι βουλευτέ. Εδώ προσοχή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό να γίνει ένα ε, παιχνίδι που να ρίχνει τις ευθύνες ε, η Κομισιόν στην Ολομέλεια και τούμπαλη. Μπορούν οι πολιτικές ομάδες να ζητήσουν απαρεξέταση ή κάποιος αριθμός βουλευτών. Και τι θα σημάνει αυτό. Θα σημάνει συζήτηση στην Ολομέλεια, επαναπομπή στην αρμόδια επιτροπή Πώς μεταφράζεται αυτή η επανεξέταση πρακτικά. Έχουμε μια εντολή, την οποία έχει εγκρίνει ας πούμε η παρούσα επιτροπή δική μας και λέει στους διαπραγματευτές, κύριοι, ορίστε, αυτή είναι η στόχη και πηγαίνετε να διαπραγματευτείτε. Αυτό ας Πώς θα το αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε τους προσανατολισμούς. Θα τους ξαναστείλουμε στην αρμόδια επιτροπή για να ξαναδούν την εντολή να κάνει πρόταση στην Ολομέλεια για να βάλει και άλλα ε, στην εντολή η Ολομέλεια. Δεν κατάλαβα. Θα πρέπει να συγκεράσουμε, είπαμε, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των βουλευτών, αλλά και την αποτελεσματικότητα, να μην την ξεχνάμε αυτή, γιατί αν τελικά η διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση είναι για να τελειώνουμε γρήγορα και ταυτόχρονα τη φορτώνουμε τόσο πολύ με μια παράλληλη διαδικασία που μας ε, υποχρεώνει να επανεξετάσουμε κάτι που έχει ήδη εξετάσει μια αρμόδια επιτροπή, θα χάσουμε το στόχο ενδεχομένω. Λοιπόν, ω εισηγητή είμαι στη διάθεσή σας και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να ακούσουμε όλες τις προτάσεις για να δούμε τελικά πού θα καταλήξουμε, γιατί αυτό έχει σημασία. Πώς θα συνδυάσουμε τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την αποτελεσματικότητα για ένα αποτέλεσμα που να μα ικανοποιεί όλου. Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Ε, το Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο χρόνος πιέζει και γίνεται όλο και λιγότερος όσον αφορά το θέμα που προχωρεί προς ψήφιση και έγκριση. Το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος τώρα και δεν θα προσπαθήσω όλα τα προβλήματα να τα θίξω και να τα καλύψω αυτά που βλέπω να υφίστανται, αλλά μόνο τις ουσιοδέστερες γραμμές. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η έκθεση πρέπει να συζητηθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και βάθος στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή διότι θα έπρεπε να στοχεύουμε οπωσδήποτε σημαντικά θέματα, να μην τα ψηφίσουμε με επίμαχο τρόπο και τριβές, αλλά να υπάρχει συνένεση σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Από πλευράς μου ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γερέρο για το έργο που έχει επιτελέσει για αυτά τα θέματα. Είναι ένα πολύ περίπλοκο σύνολο ζητημάτων και πρέπει σε βάθος να, το επεξεργαστούμε, να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά. Ένα θέμα μόνο θα ήθελα σύντομα να αναφέρω και να καλύψω. Κάνουμε εδώ λόγο για μια διαδικασία που εμείς σε επίσημε αποφάσεις και τυπικέ επίσημε αποφάσεις για μελλοντικού κανονισμούς, οδηγίες και τα λοιπά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα προβαίνουμε σε διαπραγματεύσεις προ έγκριση. Εδώ διαπραγματεύεται κάποιο και δεν διαπραγματεύεται για λογαριασμό του αλλά για το σύνολο του Κοινοβουλίου. Δηλαδή διαπραγματεύεται το σύνολο του Κοινοβουλίου, το Ευρωκοινοβούλιο. Και εδώ ακριβώς για αυτή την εντολή πρόκειται, εντολή διαπραγματευτική και για την ακόλουθη διαδικασία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την απόφαση για την αξιολόγηση αυτών με τέτοιο τρόπο ώστε συνολικά πραγματικά το Ευρωκοινοβούλιο σύνολο να μπορεί να δρά και να εκπροσωπείται. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι μια εντολή από πλευράς του συνόλου του Ευρωκοινοβουλίου απαιτείται για αυτή τη διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει ότι στην Ολομέλεια τροποποιήσεις, ε, τροπολογίες για μια τέτοια εντολή, για μια τέτοια διαπραγμάτευση πρέπει να είναι εφικτές με την παραδοσιακή ε, καλή αποτελεσματική μορφή ώστε να μπορεί αυτό να τροποποιεί την ε, εντολή ώστε στο τέλος να υπάρχει η αποκριστάλωση της, του και ψηφίσματος επ' αυτού. Από την άλλη πλευρά έχω την ανησυχία ότι κάποιες διατυπώσεις δεν είναι αρκετά σαφείς ε, και αρκετά διαφανής. Λέγεται ότι ο διοντολογικός κώδικας θα εφαρμόζεται όσο είναι εφικτό και σκόπιμο, as far as appropriate. Δεν μου φαίνεται ότι αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό για την επίλυση των προβλημάτων. Τα αποτελέσματα είναι το ουσιαστικό και δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε ότι η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και η ολομέλεια του κοινοβουλίου θα πρέπει να αξιολογούν διαδοχικά αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτό δεν μπορεί να επαφήνεται σε μια μικρή ομάδα διαπραγματευτική. Είτε είναι οι συντονιστές, είτε είναι οι ε, σκιώδεις, οι και οι συντονιστές. Είναι ένα θέμα όπου το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και μετά το σύνολο της Ολομέλειας θα πρέπει να ψηφίζουν και να εγκρίνουν. Και έτσι ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο τονίστηκε και από τη διάσκεψη των Προέδρων. Τώρα δεν είναι η χρονική στιγμή πλέον να τα συζητήσουμε όλα αυτά σε βάθος ε, σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση για υστερότερη στιγμή. Όμως στόχος πρέπει να είναι να καταλήξουμε σε μια καθαρή, διαφανή διαδικασία που θα είναι αποτελεσματική και λειτουργική και θα μπορεί από όλους να υποστηρίζεται ώστε το σύνολο του Κοινοβουλίου να μπορεί να αποδίεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε, δεν θέλω αν θέλετε να σχολιάσετε, αν πιστεύετε ότι είναι όριμη γενικά η συζήτηση έτσι ώστε να ακούσουμε κάποια από τα τελευταία σχόλια, για τα τελευταία σχόλια. Εν πάση περιπτώσει, ε, σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά περιμένουμε την άποψη. Ο κύριος Γερέρο, μάλιστα, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν και που εκφράστηκαν ε, απόψει τονίζοντα κάποια από τα θέματα που ακόμα μπορεί να εξακολουθούν να είναι προβληματικά μέσα στο πλαίσιο αυτή τη έκθεση. Θέλω να ξεκινήσω υπενθυμίζοντα κάτι. Αυτό το το οποίο επεσήμανε ο κύριος Μέντεφ Τεβίγο. Δηλαδή τελικά στο τέλος τέλος η απόφαση, η απόφαση λαμβάνεται από το κοινοβούλιο πάντα. Δηλαδή για τη συζήτηση, για το αν η απόφαση λαμβάνεται ή θα λαμβάνεται ή αν η Ολομέλεια θα είναι αρμόδια. Αυτό είναι μια τεχνητή συζήτηση. Οποιαδήποτε συμφωνία επιτυγχάνεται σε μια διαπραγματευτική διαδικασία τελικά ψηφίζεται προς έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Με τρόπο ώστε εδώ περί εκείνου που πρόκειται είναι η διοργάνωση των εργασιών, ώστε αυτή η ψήφιση από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να μην γίνεται σε γενικούς όρους και εν κενό και χωρίς πληροφόρηση και ενημέρωση σε σχέση με τους ευρωβουλευτές, αλλά σαν αποκορύφωση και επιστέγασμα μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει δίνοντας, διαχέοντας αυτές τις πληροφορίες και στο τέλος ε, ε, προς έγκριση από την Ολομέλεια. Δανιέλα, παρακαλώ, Ντανιέλα. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούστηκε. Λοιπόν, θα αναφερθώ τώρα σε κάποια από τα συγκεκριμένα ξεχωριστά θέματα που τέθηκαν. Θα ήθελα όμως μια γενική, γενικού χαρακτήρα παρατήρηση να κάνω πρώτα. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο παγκόσμια όπου όλα συνολικά τα θέματα συλλήβδη να πρέπει να εγκρίνονται στην Ολομέλεια προτού ξεκινήσει η διαπραγμάτευση μια διαπραγμάτευση σε αυτή την περίπτωση με το Συμβούλιο και σε άλλη περίπτωση να πούμε μα αυτό τότε δεν είναι κοινοβούλιο, είναι άλλο πράγμα. Ε, τα κοινοβούλια έχουν κοινοβουλευτικές επιτροπές γιατί διαφορετικά δεν θα χρειαζόντουσαν τέτοιες κοινοβουλευτικές επιτροπές δεν θα χρειαζόταν να έχουμε προέδρους των σύνοδων των προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ούτε προέδρους ε, ομάδων, αλλά όλα θα ενεγράφονται στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της Ολομέλειας, της επόμενης Ολομέλειας, επερχόμενης Ολομέλειας. Και οποιοδήποτε βουλευτής θα μπορούσε να θέσει οποιαδήποτε τροπολογία και όλοι θα συμμετείχαν σε μια συζήτηση επί παντός του επιστητού. Αυτό δεν είναι κοινόβουλιο, είναι κάτι άλλο στο τέλος τέλος. Εδώ λοιπόν περί του οποίου πρόκειται ο στόχος είναι η διοργάνωση των εργασιών που με κανένα τρόπο δεν θα μειώνει ή δεν θα υπονομεύει το γεγονός ότι θα είναι το ίδιο συνολικά το Κοινοβούλιο το οποίο θα ψηφίζει και θα εγκρίνει. Τώρα, απαντώντας σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έγιναν πιο πριν, από πλευρά του διοντολογικού κώδικα, πράγματι διατηρείται εν ζωή και εξακολουθεί εδώ να υφίσταται και μεταφέρεται ένα μέρος στον κανονισμό προς εκτέλεση και συμμόρφωση. Η απόφαση για το ποιος θα συμμετέχει στην Επιτροπή τη διαπραγματευτική είναι θέμα της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ε, με εξειδικευμένο τρόπο προσδιορίζοντας τα άτομα με το όνομα και το επώνυμό τους κτλ. Και για το γεγονός ότι θα μεταφράζεται και θα λέγεται ρητά ότι θα υπάρχει μετάφραση αυτό αφορά περισσότερο τη χρονική αλληλουχία και όχι τόσο τα δικαιώματα διότι επ' αυτού όλα, όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν δικαίωμα να έχουν στη δική τους γλώσσα τα κείμενα και επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας ένα θέμα που προηγούμενα δεν θα έχει μετάφραση επί των κειμένων που, είναι, ε, που άπλονται αυτού του θέματος ε, στις άλλες γλώσσες ώστε να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να έχουν, ε, να έχουν εξοικειωθεί οι ευρωβουλευτές περί τίνος πρόκειται. Εδώ, όμως εδώ στη συνέχεια νομίζω υπάρχει κάποια μικρή σύγχυση. Ίσως δεν τα επεξήγησα εγώ καλά για το ρόλο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και τον ρόλο της διαπραγματευτικής ομάδας και των συντονιστών ισχυωδών εισηγητών. Προσέξτε, η διαπραγματευτική ομάδα όπως πολύ σωστά ανέφερε ο προλαλή σα στην παρέμβασή του, η διαπραγματευτική ομάδα εκπροσωπεί το θεσμικό μας όργανο. Σε αυτή την περίπτωση εκπροσωπεί την αρμόδια καθήλυν κοινοβουλευτική επιτροπή για το θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δίνεται η πρωτοκαθεδρία και διεύθυνση των εργασιών επ' αυτού του θέματος στον πρόεδρο της αρμόδιας καθήλυν κοινοβουλευτικής επιτροπής, διότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να επομίζεται αυτού του καθήκοντος ως υπεύθυνο και σε όλη τη διαδικασία ενημέρωσης και πληροφόρησης προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα δίνεται η πληροφορία, θα δίνονται αυτές οι πληροφορίες στο σύνολο των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που πάλι στο σύνολο της από πλευράς της θα πρέπει να ψηφίζει προς έγκριση τη συμφωνία που θα έχει επιτευχθεί από την διαπραγματευτική ομάδα. Ο γενικός κανόνας είναι πάντα λοιπόν ότι το σύνολο των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ενημερώνεται, πληροφορείται και είναι το σύνολο των μελών των Ευρωβουλευτών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που εγκρίνει απορρίπτει την επιτευχή σας συμφωνία. Και Υπάρχει και η δυνατότητα που έχουμε εξετάζεται ότι σε όλες τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών να να μπορεί να εγγραφεί ένα ε, σημείο στην ημερήσια διάταξη, αρχικό σημείο όπως στις ανακοινώσεις του Προέδρου για παράδειγμα, όπου θα ενημερώνονται τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το πώς έχει εξελιχθεί, πώς μετεξελίσσεται ένα θέμα το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και στο οποίο εμπλέκεται η Κοινοβουλευτική αυτή Επιτροπή. Μόνο κατ' εξαίρεση και για λόγους που φυσικά μπορούν ε, να ε, προσδιορίζονται κατά λεπτός περαιτέρω ή μόνο όταν υπάρχει κάποια αδιαφυσβήτητη επίγουσα περίπτωση ή σε σχέση με την ενημέρωση από τη διαπραγματευτική ομάδα προς συντονιστές ισκιώδης εισηγητές ε, ή τον πρόεδρο της Επιτροπής, μόνο τότε μπορεί να εγκριθεί αυτή η συμφωνία υποδιαπραγμάτευση που στο τέλος τέλος θα πρέπει να εγκριθεί, απορριφθεί από την ολομέλεια του σώματος. Δηλαδή δεν αφαιρείται, δεν μειώνεται το δικαίωμα, δεν συρρυκνώνεται το δικαίωμα αυτό όσον αφορά την ολομέλεια του σώματος με κανένα τρόπο. Και συμφωνώ ότι από κοινού με τους ε, συντονιστές θα πρέπει να ενημερώνονται οι σκιώδεις εισηγητές. Αυτό δεν είναι πρόβλημα καθόλου και νομίζω ότι θα άξιζε να προβληματιστούμε όπως ε, επεσήμανε ο κύριος Νταφ να αναφέρεται ρητά και να λέγεται ότι αποκλείονται οι άτυπες επαφές διότι επ' αυτού θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα σημείο το οποίο παραμένει ενισχύει στους κανόνες τους ε, δεοντολογικούς ε, και δεν υπάρχει κάποιος λόγος εδώ να ε, περάσει στο, ως θέμα κανονισμού για την κυρία Γιαννάκου και για την ε, ε, συνάντηση που ε, είχαμε και αναφέρθηκε στο ρόλο της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και πρέπει να επισημάνω ότι είμαι φυσικά ανοιχτός και πρόθυμος να δω οποιαδήποτε πρόταση για την ε, διάσκεψη των Προέδρων ή μέσω των κοινοβουλευτικών ομάδων ή μέσω αριθμού Ευρωβουλευτών να μπορεί επίσης αυτό το θέμα να τεθεί στην Ολομέλεια. Και συμφωνώ με αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Μέντες Τεβίγκο ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί η Ολομέλεια ε, να μην ξεκινά να συζητά κάθε ένα από αυτά τα θέματα της διαπραγματευτικής εντολής ε, και να ξαναρχίζει το παιχνίδι από μηδενικό σημείο και επίσης για το θέμα το οποίο την ερώτηση, το ζήτημα το οποίο έθεσε ο πρόεδρος ε, και ανέφερε και ευρωβουλευτής συμπίπτω και εγώ σε αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντική συνένεση από την ταχεία διεκπαιρέωση στην αντιμετώπιση και επίλυση αυτών των ε, θεμάτων. Και αν για να επιτευχθεί συνένεση είναι αναγκαίο στην επερχόμενη συνεδρίαση της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αντί να συζητηθούν οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τις ομάδες να επανεξεταστεί αυτό το θέμα και να ανοίξουμε μια περίοδο κατάθεσης τροπολογιών επ' αυτού δεν έχω κανένα πρόβλημα πρέπει να πω να αποδεχτώ αυτή την προσέγγιση, αυτή την πρόταση. Γι' αυτό αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. dürfte ich Κύριε Σχέφνερ, να προτείνω κάτι σε άλλα σημαντικά νομοθετήματα και διαδικασίες. Έχουμε επίσημη συζήτηση και τυπική με τους κοιόδης συγητές. Και μεταξύ μας μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα για να μην έρχονται όλα από την αρχή στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Non ho sentito niente perché non ha funzionato l'interpretazione, non so come mai. Δεν ξέρω, έχω κάποια τεχνικά προβλήματα με τη διαρμηνία, λέει ο πρόεδρος. Μπορείτε να επαναλάβετε από την αρχή. Στα αγγλικά, κύριο Σχέφνερ, για την προετοιμασία της επόμενης συνεδρίασης να έχουμε μια επίσημη συνάντηση του εισηγητού με τους Σκιώδης για να προετοιμάσουμε τη συζήτηση ακριβώς. Αλλιώς θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή στην Ολομέλεια της Επιτροπής αυτή τη συζήτηση. Ε, θα δούμε, δεν ξέρω τι πιστεύει ο εισηγητή. είναι ελεύθερο να προτείνει την μέθοδο που θα ακολουθηθεί η συζήτηση, μπορούμε να μην καθορίσουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών στην παρούσα φάση. Εγώ προσωπικά βέβαια εκτιμώ ότι το επίπεδο της συζήτηση έχει οριμάσει αρκετά. Το μοναδικό θέμα είναι το πόσο θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στην, στον έλεγχο των διαπιστευτηρίων από την Ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας κυνηγάει χρονικά, δεν καθορίζουμε προθεσμία κατάθεσης τροπολογίας, ο εισηγητής θα συναντηθεί εκ νέου με τους σκιώδεις εισηγητές και θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνάντηση. Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ τώρα πλέον τις ψηφοφορίες. Ξεκινώντας, έχουμε την έκθεση για την τροποποίηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 για τις πρωτοβουλίες των πολιτών, την πρωτοβουλία των πολιτών δηλαδή η έκθεση του κυρίου Στάνιμιρ Ήλτσεφ. Δεν ξέρω αν θέλετε να παρουσιάσετε την σύστασή σας. Κύριε Ήλτσεφ, θέλετε το λόγο. Όχι, λέει ο κύριος Ήλτσεφ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε σε ψηφοφορία. Θέτω σε ψηφοφορία καταρχάς. Δεν θέλει κανείς άλλος τον λόγο, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος, μπορούμε να ψηφίσουμε. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 2 Χέφνερ. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Ποιος είναι υπέρ της 2. Κατά της 2. Ποιος απέχει, απορρίπτεται προφανώς η 2. Τροπολογία 1 του ιδίου του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται και οι δύο. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα. Η 3 ήταν ταυτόσιμη με την 1 οπότε δεν την ξαναψηφίζουμε. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της τροπολογίας 4. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή ομόφωνα. Τροπολογία 6 είναι υπέρ. Κατά. Ναι, αποχές δύο, κατά και οι υπόλοιποι υπέρ, δεκτή η 6. Ψηφίζουμε τώρα πλέον το σύνολο της πρότασης. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκαεννέα υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ένας κατά. Ποιος απέχει. Μία αποχή. Γίνεται λοιπόν δεκτή η έκθεση αυτή. Συγχαρητήρια κύριε Ήλτσεφ. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Αφορά την έκθεση του 2010. Η κυρία Γκουρμάη, η οποία δεν είναι παρούσα βέβαια η κυρία Γκουρμάη, γιατί ασχολείται με την ισομερή συνέλευση ΑΚΕ. Αλλά αντικαθίσταται από τον κύριο Γκουερέρο, ο οποίος έχει το λόγο εφόσον θεωρεί ότι είναι χρήσιμο. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο, δεν είναι απαραίτητο να μιλήσω. Εγώ το είπα αυτό, απλά δικαιολογώντας την απουσία της συναδέλφου Τσιταγκούρμαϊ αλλά έχουμε τον κύριο Γκουερέρο εδώ, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα του στην ψηφοφορία. Δεν θέλετε το λόγο λοιπόν κύριε Γκουερέρο. Συνεχίζει χωρίς μικρόφωνο, ο πρόεδρος δεν τον ακούμε. Α, ναι, ξέχασα. Λοιπόν, θέτω σε ψηφοφορία την ένα Γκριπ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Γίνεται δεκτή η τροπολογία Λεγκρίπ. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία Πάξας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η έξι Μέλτσα. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 4 έχω πάντα την τροπολογία 3 του κυρίου Νταφ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στην τροπολογία 10 έχω μια προφορική τροπολογία. Την γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας τη διαβάσω. Α, για μια στιγμή κάτι ξέχασα, δεν φτάσαμε στη 10, λέει ο πρόεδρος, το συγγνώμη, πάω πίσω. Έχουμε την τροπολογία 5 της κυρίας Γιαννάκου, ποιοι είναι υπέρ. Αποχές. Α, ναι, κατά έπρεπε να πω, συγγνώμη. λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Και è contrario? Κατά. Αποχές. Δεκτή η τροπολογία ακού. Τροπολογία 4 Λεγκρίπ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Τέσσερις κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 7. Κυρία Γιαννάκου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9. Ήλτσεφ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Φτάσαμε τώρα επιτέλους στην 10. Εδώ υπάρχει μια προφορική συμπλήρωση τροπολογία, την οποία γνωρίζετε, υπάρχει γραπτά έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Κυρία Λεγκρίπ, ναι, ε, εσείς θέλετε αν, να πούμε αν δεχόμαστε με το να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Ναι, ναι, ερμηνεύσατε πάρα πολύ σωστά λέει ο Πρόεδρος, εκτατικά ερμηνεύσατε θα έλεγα ε, την ερώτηση την οποία σας έκανα. Έπρεπε να κάνω διαφορετικά την ερώτηση. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε αν κάποιος είναι εναντίον αυτής της προφορικής τροπολογίας γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα η ψηφοφορία. Είστε πολύ λογικός άνθρωπος κυρία Λεγκρίπ, οπότε δεν θα δεχθούμε την προφορική τροπολογία, δεν τη θέτω σε ψηφοφορία, θέτω όμως σε ψηφοφορία την τροπολογία 10 Ιλτσεβ, ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή, ποιοι είναι κατά, α, α, ένας είναι κατά. Αποχές δεκτή. Λοιπόν, τροπολογία 11, Ήλτσεφ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Λοιπόν, δεν γίνεται δεκτή. Τροπολογία 12, Άντζιου Ντάφ, ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. τροπολογείο 13. η Ήλτσεβ. Είναι υπέρ. Κατά. απορρίπτεται. Τροπολογείο 14 στην παράγραφο 7 Ήλτσεφ και είναι υπέρ. Λοιπόν, δεκτή η προηγούμενη τροπολογία. Ψηφίσουμε την 15 Νταφ. Ποιοι είναι υπέρ. κατά απορρίπτεται. Δεκαέξι πάξας, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Δεκαεπτά μέλτσα, ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18 DAF ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 Ήλτσεφ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 20 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή Φτάσαμε τώρα στη συμβιβαστική τροπολογία, τη μοναδική συμβιβαστική τροπολογία, την οποία καταθέτει ο εισήγητης στην παράγραφο 10. Είναι υπέρ. Λοιπόν, συμβιβαστική στην 10 ψηφίζουμε. Κατά. Απορρίπτεται η συμβιβαστική. Ψηφίζουμε τώρα τις επόμενες τροπολογίες, τις οποίες ήθελε η συμβιβαστική να συμπεριλάβει. Λοιπόν, 21 της κυρίας Λεγκρίπ, ποιοι είναι υπέρ. 24. Α, για μια στιγμή, για μια στιγμή. Λοιπόν, ε, είδαμε ε, τους υπέρ ε, της 21 Λεγκρίπ. Ποιοι είναι κατά. Ποιος απέχει. Δεκτή. Α, η 21. έχει καταπέσει 24, έχει καταπέσει 22, έχει καταπέσει 25 μέλτσα, όπως και 23 Χέφνερ. Φτάνουμε τώρα στην τροπολογία 26 Ιλτσεφ. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 DAF ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 DAF ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 29 λεγκρίπ ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές δεκτή. Η 30 Χέφνερ ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 Γκουερέρο υπέρ. κατά αποχές δεκτή. 32 λεγκρίπ, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 34 της κυρίας Γιαννάκου υπέρ. Α, για μια στιγμή η κυρία Λεγκρίπ έχει ζητήσει το λόγο. Συγγνώμη που διακόπτω την ροή των ψηφοφοριών. Θα ήθελα όμως μια μικρή διευκρίνηση σημασιολογικού ίσως τύπου Ίσως να τίθεται ένα θέμα μετάφρασης εδώ, αλλά στο γαλλικό κείμενο της συγκεκριμένης τροπολογίας χρησιμοποιείται η λέξη εθνικότητα, αλλά στα αγγλικά η λέξη nationalité, συγγνώμη, στα γαλλικά και στα αγγλικά η λέξη citizenship. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αναφέρεστε στην 34 της κυρίας Γιαννάκου. Το πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα. Η κυρία Γιαννάκου θα πρέπει να μας πει ακριβώς τι θα πρέπει να προτιμήσουμε. Γένεια. Λοιπόν, η Allora, αυτή είναι η σωστή η λέξη της κυρίας Γιαννάκου, citizenship. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 34, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή η τροπολογία 33 της κυρίας Λεγκρίπε ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή μπορούμε λοιπόν τώρα να ψηφίσουμε στην τροπολογημένη πρόταση ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές λοιπόν δεκτή 17 υπέρ 3 ε, κατά συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή θα πρέπει τώρα να περάσουμε στην τελευταία ψηφοφορία η έκθεση Ρέγνερ ο κύριος Γουερέρο παίρνει το λόγο ναι κύριε Πρόεδρε Εχθές στη συνεδρίαση των συντονιστών, ετέθη ένα ζήτημα. Θεωρήθηκε σκόπιμο να ζητήσουμε, να συμβουλευτούμε την νομική υπηρεσία για τις ερωτήσεις που έκανε ε, η συγγήτρια και ο κύριος Χέφνερ και ο κύριος Μέντες Δεβίγο. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ψηφίσουμε την γνωμοδότηση πριν ψηφίσει η καθήλυνα αρμόδια νομική επιτροπή στην οποία γνωμοδοτούμε. Δυστυχώς τώρα απουσιάζει και η συντάκτρια της γνωμοδότησης αυτή τη στιγμή, η οποία κανονικά θα είχε δικαίωμα να ζητήσει να ψηφιστεί η γνωμοδότησή της, μια που είναι στην ημερήσια διάταξη. Αλλά εάν υπάρχει πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής που ε, θεωρεί σκόπιμο να μην ψηφιστεί, να αναβληθεί και να βρεθεί κάποια στιγμή στο Στρασβούργο για να ψηφίσουμε ειδικά αυτό το θέμα, η πολιτική μου ομάδα θα ήταν διατεθειμένη να το δεχτεί. Δηλαδή, δύο τινά, είτε ψηφίζουμε σήμερα και ε, διαβιβάζουμε τη γνωμοδότησή μας μαζί με την άποψη της ε, νομικής υπηρεσίας είτε θα βρούμε μια στιγμή στο Στρασβούργο για να ψηφίσουμε όταν θα έχει γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία και πριν ψηφίσει η νομική επιτροπή. Εντάξει. Ο κύριος Νταφ. Πρόεδρε, συμφωνώ με την αναβολή της ψηφοφορίας για το θέμα αυτό, ιδιαίτερα απουσία της συντάκτριας της νομοδότησης. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία μεταξύ των νομικών και της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την πρόταση αυτή. Ειλικρινά δεν έχουμε συζητήσει το θέμα στην ουσία του, στην Επιτροπή μας. Το προηγούμενο είναι άκρο σημαντικό, διότι ιδρύουμε ένα είδος εφετείου στο δικαστήριο. για τη συμφωνία ε, για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που δεν είναι τμήμα του κοινοτικού δικαίου. Ακριβώς επειδή το θέμα είναι τόσο περίπλοκο όσο και σημαντικό, πιστεύω ότι χρειάζεται αναβολή αν θέλουμε να αποφασίσουμε έτσι, με σοβαρότητα και παρουσία της εισηγητρίας και να ακολουθήσουμε και τη συμβουλή της νομικής μας υπηρεσίας. Ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε και από την Νομική Επιτροπή να αναβάλει και εκείνη την ψηφοφορία της. Στις 20 Δεκεμβρίου προβλέπεται να ψηφίσουν. Μπορούμε να ζητήσουμε να ψηφίσουν τον Ιανουάριο για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ναι, Πρόεδρε, συμφωνώ με αυτά που είπε ε, και ο, ο εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών και των Φιλελευθέρων. Δεν έχει νόημα να ψηφίσουμε αφού λείπει και η κυρία ε, Ρέγνερ, αλλά για να είμαστε συνεπεί με τα όσα αποφασίσαμε εμεί στο Λαϊκό Κόμμα, θα θέλαμε η γνωμοδότηση οπωσδήποτε να ψηφιστεί πριν την έκθεση τη Νομική Επιτροπή. Αυτό που λέει ο κύριο Δάφη έχει αρκετό νόημα. Θα μπορούσατε, κύριε Πρόεδρε, σα παρακαλώ, να μιλήσετε με τον κύριο Λένα και να του ζητήσετε να το αναβάλει μέχρι το Γενάρη. Δεν χάλασε και ο κόσμο. Ε, αντί για τι 20 Δεκεμβρίου. Αλλιώ να ζητήσουμε έκτακτη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της ε, συνόδου στο Στρασβούργο ακριβώς για αυτό το θέμα, για να γνωμοδοτήσουμε. Είναι σημαντική η γνωμοδότησή μας και πρέπει να υπάρχει. Κατά τα άλλα συμφωνώ και με τον κύριο Γκερέρο και τον κύριο Ντάφ. Εφνερ. Ναι, Στο τέλος, τέλος συμφωνώ και εγώ με αυτή την πρόταση. Αυτή τη στιγμή πιστεύω δεν μένει τίποτα άλλο πια παρά αυτό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να εκφράσω και την έκπληξή μου. Αμέσως όταν μας διαβιβάστηκε αυτό, αποσαφηνήσαμε ότι εδώ έχουμε σημαντικές νομικές επιφυλάξεις και ζητήσαμε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Είχαμε πολυάριθμες συζητήσεις με την κυρία εισηγήτρια επ' αυτών. Δεν πρόκειται εδώ για ένα θέμα στο περιθώριο και επουσιώδες, αλλά για το κύριο, κέριο θέμα. Τι θα κάνουμε εμείς ως Συνταγματική Επιτροπή και πώς θα τοποθετηθούμε στα άλλα θέματα, αν στο πιο αποφασιστικό θέμα δεν έχουμε σαφήνεια. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά για να μην ε, αυτογελιοποιηθούμε, θα πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί. Θέλω επίσης να εκφράσω την εκπληξή μου για το ότι σύμφωνα με τα σαφή θέματα και αμφιβολίες που υπάρχουν, η εισηγήτρια σήμερα προφανώς θεωρεί ότι μπορεί να ψηφιστεί η έκθεσή της χωρίς η ίδια να συμμετέχει. Δεν νομίζω ότι έτσι μπορούμε να διαβουλευτούμε από αυτών των θεμάτων και θα πρέπει να αναμείνουμε τη γνωμοδότηση της νομικής μας επιτροπής και να πούμε στην εισηγήτρια ότι θα μας ευχαριστούσε αν στις 20 τόσες του μήνα θα μπορούσε να συμμετάσχει και να συζητήσει και μαζί μας για αυτά τα θέματα, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Γκερέρο ζήτησε πάλι να παρέμβει, παρακαλώ. Να τα πάρουμε με τη σειρά, Πρόεδρε. Νομίζω ότι επαρκώς είναι πλέον σαφές, αλλά θέλω να το επαναλάβω για άλλη μια φορά εγώ. Δηλαδή με άλλα λόγια. Εμείς ε, χρονικά εξαρτώμεθα από την απόφαση της νομικής επιτροπής που είναι η καθήλυνα αρμόδια. Επί της ουσίας είμαστε σε σχέση με την έκθεση, τη γνωμοδότηση της νομικής μας επιτροπής εξαρτώμαστε από αυτήν. Όμως ο χρόνος είναι το σημείο κλειδί, το πιο σημαντικό στοιχείο. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε χωρίς να υπάρξει μια ε, για την ουσία επί της νομικής επιτροπής τοποθέτηση χωρίς να έχουμε την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε δικαίωμα να γνωμοδοτήσουμε αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Και όπως επεσήμανε ο κύριος Μέντες Δεβίγο, αν ε, ε, η Υπηρεσία Νομικών Υποθέσεων αναβάλει την ψηφοφορία της και εμείς θα μπορούσαμε να αναβάλουμε τη δική μας. Όμως ε, καθώς η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αν αποφασίσει να ψηφίσει παρόλα αυτά στις 20 Δεκεμβρίου τότε εμείς με ή χωρίς τη γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών θα έπρεπε να ψηφίσουμε πριν από τις 20 υποχρεωτικά και αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο κάποτε στο Στρασβούργο, στην Ολομέλειά μας. Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπε μόλις τώρα ο κύριος Γκουερέρο εκφράζει όλα όσα πιστεύουμε. Υπάρχει μια συνένεση από ό,τι φαίνεται. Θα έρθω σε επαφή εγώ για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα αναβολής λοιπόν στη νομική επιτροπή και αν δεν γίνεται αυτό ίσως να ζητήσουμε μία έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής μας την Δευτέρα του Στρασβούργου. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Ίσως εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία αντιστροφή στην ημερησία διάταξη και να συζητήσουμε το θέμα της τροποποίησης του κανονισμού στις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο και το Eurogroup. Ο εισηγητής, ο κύριος Λαμασούρ, μας είπε ότι μπορεί να είναι εδώ μέχρι τις 11.30 γιατί έχει άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις, οπότε νομίζω ότι οφείλουμε και εμείς να έλθουμε τώρα πλέον στη συζήτηση αυτή με τον κύριο Λαμασούρ. Ζητήθηκε η έκθεση αυτή από τη διάσκεψη των Προέδρων, θυμίζω, για να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο τη νέα θεσμική και συνταγματική ισορροπία ανάμεσα στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και θα πρέπει η έκθεση αυτή να ασχοληθεί ε, με τα θέματα τα οποία εμείς θέλουμε προς εξέταση και τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις διακανονιστικού τύπου. Θα δώσω λοιπόν πρώτα τον λόγο στον συνάδελφο Λαμασούρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω φτιάξει ένα μικρό έγγραφο εργασία για να δούμε πώς έχει η κατάσταση δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, συνόλου του Συμβουλίου. ενώ όλα τα θεσμικά ε, όργανα που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Σκέτο που είναι Συμβούλιο Υπουργών και ε, πιο κάτω κορεπέρ, ομάδε εργασίας και πάει λέγοντας. Δύο χρόνια λοιπόν αργότερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο ικανοποιητική και ότι η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν γίνεται αισθητή ως θα όφιλε. Για να μην πω ότι έχει μειωθεί και η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες του Συμβουλίου. Προσθέτω δε ότι σε σχέση με τη στιγμή που εκπώνησα το έγγραφο αυτό, έχουν επιταχυνθεί εξελίξεις. Και σήμερα όλο και πιο συχνά ακούμε φωνές στην Ευρώπη να ζητούν νέα συνθήκη. Και θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια γι' αυτό. Γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ ε, σοβαρή, αυτή που διανύει σήμερα η Ευρώπη, και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τη συνθήκη της Σαββόνας, για τις ενδεχόμενες ανεπάρκειές της, αν χρειάζεται συμπλήρωση ή ακόμα και αναθεώρηση. Πώς λοιπόν έχουν σήμερα τα πράγματα. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει κάνει θεσμικό όργανο, ένα όργανο που ήδη υπήρχε, που ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και του έχει δώσει και ένα πρόεδρο Και ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συνθήκε είναι να ορίζει τις μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές και τους προσανατολισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που ίσχυε και από το παρελθόν, και να συντονίζει τις εθνικές πολιτικές σε τομείς όπου η αρμοδιότητα παραμένει ουσιαστικά εκείνη των κρατών μελών, αλλά όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη νομική υποχρέωση μέσω της Συνδίκης Λισαβόνας αλλά και την πολιτική υποχρέωση για λόγους αποτελεσματικότητας να συντονίζεται. Οπότε αυτός ο συντονισμός γίνεται με τρόπο πάρα πολύ λογικό από τους Πρωθυπουργού, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κλπ. Τι διαπιστώσαμε λοιπόν. Ακριβώς και λόγω της κρίσης και όχι μόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει λόγω της κρίσης ή των κρίσεων που συγκλονίζουν από το 2008 την Ένωση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανειλημμένα συνεδριάζει. Και de facto γίνεται ένα είδος συλλογικής εκτελεστικής εξουσίας σε τομείς που αυξάνονται συνεχώς. Και ορισμένοι έχουν κοινοτική αρμοδιότητα και θα έρθω σε αυτό, αλλά πιο συχνά είναι τομείς που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και βγαίνουν από το συντονισμό τον αμυγή της ε, πολιτικής σε κοινωτικό επίπεδο. Αυτό όμως πλέον ε, είναι πρόβλημα για το Κοινοβούλιο. Γιατί το Κοινοβούλιο στην νομοθετική του εργασία έχει ως συνομιλητή αποκλειστικό το Συμβούλιο Υπουργών. Αλλά από ό,τι φαίνεται σε όλα τα σοβαρά ζητήματα και τα σπουδαία, οι πραγματικέ αποφάσει, οι πολιτικέ αποφάσει, εντάξει νομικά είναι το Συμβούλιο Υπουργών, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις ε, που έρχεται να εκτελέσει το Συμβούλιο Υπουργών λαμβάνονται πλέον σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αν θέλει το Κοινοβούλιο εγκαίρως να επεμβαίνει εκ των προτέρων για να λαμβάνονται υπόψη ανησυχίε του, οι απόψει του, οι θέσει του από τα όργανα που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ανταλλάσσει απόψεις, αν μη τι άλλο, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όχι να διαπραγματεύεται, γιατί αυτό δεν είναι ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα των θεσμικών οργάνων. Αλλά να ανταλλάσσουμε απόψει, να έχουμε κάποια επαφή. Έχουμε μεγάλε δυσκολίε για να το πραγματοποιήσουμε αυτό για θέματα πολύ διαφορετικά όπως είναι το σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, η ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχία, όλα αυτά αποφασίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και το Κοινοβούλιο έρχεται να επέμβει μόνο στο στάδιο της νομικής υλοποίησης χωρίς να έχει την επιρροή που θα όφιλε εκ των προτέρων σε αυτά τα θέματα. Έρχομαι τώρα στα δημοσιονομικά προβλήματα που γνωρίζω καλύτερα γιατί είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Πέρυσι είχα την εξή δυσκολία, την οποία ξεπεράσαμε τελικά, αλλά με όρους που δεν μας ικανοποιούν από πλευράς ε, διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως το ψήφισε το Συμβούλιο, που ήταν μέγας συμβιβασμό και μεγάλη υποχώρηση που δεν είχε κάνει ποτέ το Κοινοβούλιο. Πρότεινε λοιπόν το Κοινοβούλιο σε αντάλλαγμα μια πολιτική συμφωνία για να συνεργαζόμαστε καλύτερα τα δύο θεσμικά όργανα για να προετοιμάζουμε το νο... δημοσιονομικο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Χρειαζόταν δηλαδή πολιτική συμφωνία για να συμπληρωθεί για τον προπολογισμό η συνδέχιση τη Το πρόβλημα λοιπόν το διαδικαστικό που διαπιστώσαμε πέρσι ποιο ήταν συνομιλητή μα ήταν οι υπουργοί αρμόδιοι για τον προπολογισμό, οι οποίοι μα είπαν Ωραία τα λέτε, αλλά εμεί εντολή έχουμε για να διαπραγματευτούμε μόνο τον προπολογισμό του 2011. Πολιτική πτυχή για τι διαδικασίε δεν είναι δική μα υπόθεση, να αποτανθείτε αλλού, αρμοδίω. Με δέχτηκε ο κύριος πάει με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια και καλοσύνη. Αποτανθήκαμε στη Βελγική τότε Προεδρία και κάναμε μια τρύπα στο νερό Τελικά βρήκαμε μια συμφωνία με την Ουγγρική Προεδρία που διαδέχτηκε τη Βελγική, η οποία δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της να ε, θεσπίσει ένα μηχανισμό που θα εγγυάται ότι κάθε φορά που το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα ασχολείται με ε, τις δημοσιονομικές προοπτικές, αμέσως πριν και αμέσως μετά θα συναντάτε με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης διαπραγματευτήκαμε στη συνέχεια με την Πολωνική Προεδρία για να το κάνει ε, και τη Δανική και τώρα διαπραγματεύομαι με την Ιρλανδική. Τελικά θα καταφέρουμε ε, να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν είναι ικανοποιητικό. Και φαντάζομαι και σε άλλους τομεί πέρα από τα ε, θέματα του προλογισμού θα έχουμε και τις ίδιες δυσκολίε. Λοιπόν, τίθεται τώρα το εξή ζήτημα για την εφαρμογή της συνθήκη Λισαβόνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ποιο τρόπο μπορεί να υλοποιήσει μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ τον πρώην συνάδελφο Ρίτσαρτ Κόρμπετς που είναι παρόν εδώ σήμερα ε, και που μας έδωσε την προσωπική του άποψη για το έγγραφο εργασίας και έκανε και κάποιες διορθώσεις. Βεβαίω το οριστικό κείμενο θα τις λάβω υπόψη μου γιατί είναι δικαιολογημένες. Ο πρόεδρος Φαν επέδειξε τεράστια προθυμία να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι και δική σας, της Επιτροπής σας, ότι οι σχέσεις μας θα πρέπει να είναι και πιο πολυάριθμες και πιο καλά οργανωμένες. Η σημερινή κατάσταση όμως δεν εξαρτάται από τη βούληση και την προθυμία του Πρόεδρου Φαρόμπαη, αλλά από τα υψηλά όργανα του Κοινοβουλίου μας, ιδιαίτερα από τη διάσκεψη των Προέδρων. Έτσι είναι κάπως λεπτό αυτό το θέμα. Δηλαδή πριν ασχοληθούμε με τους άλλους θα πρέπει να κανονίσουμε τα του οίκου μας. Και κάτι άλλο που είναι αρκετά έτσι, πώς να το πω, ενοχλητικό. Κάθε φορά που συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι συζητήσεις που γίνονται, ε, ε, πώς γίνονται. Έρχεται ο Πρωθυπουργός της ε, εκάστοτε Προεδρίας, που μας έχει κάνει και τις προγραμματικές του δηλώσεις στην αρχή του εξαμήνου, που δεν έχει κανένα νόημα, γιατί δεν είναι σε επίπεδο κυβέρνησης πια οι προγραμματικές δηλώσεις στην εκπεριτροπής Προεδρία. Στη Δανία, ας πούμε, είναι εξαίρετη πρώην συνάδελφος κυρία Τόνι Σμιτ, η γοργόνα της Κοπεχάγης που ανέλαβε τώρα πρωθυπουργό της χώρας και χαιρόμαστε όλοι που θα τη δούμε, αλλά ε, δεν μπορεί να κάνει προγραμματικέ δηλώσει τη Δανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει πια νόημα. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, έρχεται ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κ. Φαρόμπε, που μας τα εξηγεί όλα αυτά και λογοδοτεί. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται κατά με αναθεώρηση. Πανεξέταση, αν μη τι άλλο. Και επίση τίθεται και ένα πρόβλημα για την Ευρωζώνη διότι έχουμε το Eurogroup με τον μόνιμο πρόεδρο του, αλλά τώρα γίνονται και σύνοδοι κορυφή της Ευρωζώνης. Και διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται να διοργανώσουμε ένα είδο ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των συνόδων κορυφής τη Ευρωζώνης. Προσθέτω επίσης ότι η χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε τις κυβερνήσεις στο να ενισχύσουν όλα ε, τα θέματα που έχουν σχέση με τη δημοσιονομική επιθαρχία και τη συμπληρώνουν και με ένα είδος πολιτικής συμφωνίας. Διευκρινίζουν τις συνθήκες, ας πούμε, μέσω του λεγόμενου six-pack. Ξέρετε το πακέτο των έξι οδηγιών για την οικονομική διακυβέρνηση. Η δε εμπειρία έχει αποδείξει ότι Πολιτικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο στα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια και η κοινή γνώμη των κρατών να δεχθούν αποφάσεις που αφορούν το περιεχόμενο της δημοσιονομικής πολιτικής ή τους προσανατολισμούς της φορολογικής πολιτικής ή άλλης οικονομικής πολιτικής λαμβάνονται ως αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης ή της Ευρωζώνης χωρίς δημόσια συζήτηση. Μα είμαστε δημοκρατικά καθεστώτα, δημοκρατικές χώρες με παράδοση. Ό,τι έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό είναι στην καρδιά και της κυβερνητικής αλλά και της κοινοβουλευτικής ζωής. Ας πούμε η συμφωνία για την ενίσχυση και την επέκταση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 21 Ιουλίου του EFSF που είχε καταστεί κατεπίγουσα αυτή η συμφωνία λόγω της κατάστασης των αγορών, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς να έχουν εξετάσει αυτή τη συμφωνία, συζητήσει και εγκρίνει και τα 17 κοινοβούλια της Ευρωζώνης. Και χρειάστηκε πάνω από δυόμιση μήνες αυτή η ιστορία. Με τις γνωστές δυσκολίες σε κάποιες χώρες, ψυχόδραμα στη Σλοβακία που δεν δεχόταν ε, η Βουλή να κυρώσει αν δεν είχε ρίξει την κυβέρνηση. Και τελικά όταν έφτασε να εφαρμοστεί είχε καταργηθεί από τις εξελίξεις στις αγορές και αντικαταστάθηκε από μια άλλη συμφωνία της 26 και 27 Οκτωβρίου όπως ξέρετε. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά. Έχουμε και άλλο πρόβλημα τώρα, το οποίο έχει να κάνει με τις σχέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο ή τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης. Διανύουμε τώρα μια περίοδο που ερχόμαστε να διαπιστώσουμε ότι χρειάζεται κάπως να συμπληρωθεί αυτός ο μηχανισμός που έχει δημιουργηθεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας με πιο επίσημη σχέση και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με τις συνοκορυφείς της Ευρωζώνης αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια όπως επίσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να εξετάσει διάφορες προτάσεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα σας έλεγα ότι το ερώτημα που τίθεται είναι δεν θα μας συνέφερε να διαπραγματευτούμε ένα είδος συμφωνίας κυρίων που να ονομάζεται αλλιώ, δεν ξέρω. Νομικά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, διοργανική συμφωνία ή για να φτάσουμε στην άλλη άκρη ε, ισχύω από πλευρά μπορεί να είναι απλή ανταλλαγή επιστολών. Αλλά κάπω να επισημοποιηθεί αυτή η σχέση μα και η συνεργασία. Και είναι θέμα αυτό τη Επιτροπή σα, συνταγματικών υποθέσεων. Πέρα από όλα αυτά, τα προβλήματα, τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε ο κόσμος να προβληματίζεται δημόσια ε, ο κόσμος εννοώ οι αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, πρόεδροι κομμάτων στα συνέδριά τους, σε μεγάλα πολιτικά κόμματα, εκφράζονται απόψεις, μήπως χρειάζεται να συμπληρωθεί, να αναθεωρηθεί, να επανεξεταστεί η συνθήκη της Αφώνας. Και νομίζω ότι και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα πρέπει να προβληματιστεί. Αν έχει έρθει άραγε η ώρα να αποφανθεί και εκείνη. Γιατί μου κάνει εντύπωση και έκπληξη και με ανησυχεί κάπως ο τρόπος ξέρετε, που έχει γίνει αυτή η συζήτηση και η πορεία που έχει πάρει. Ε, πολύ υψηλά πολιτικά στελέχη κάνουν δηλώσεις που δείχνουν ότι δεν γνωρίζουν καλά το περιεχόμενο της συνθήκης της Λισαβόνας. Συμπεριλαμβανομένων εδώ και ορισμένων ε, υπογραφούντων της συνθήκης. Εκπλήσωμε που ε, φανίστηκε ως τρομακτική καινοτομία η εκλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με καθολική ψηφοφορία. Μα αυτή τη λέει η συνθήκη της Λισαβόνας. Εντάξει, όχι σύμφωνα με το προεδρικό, αμερικανικό ή γαλλικό πρότυπο, αλλά σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό πρότυπο, αλλά γερμανικά ή ισπανικά. Την Κυριακή, κανένας Ισπανός ψηφοφόρος δεν έριξε ψηφοδέλτιο που να γράφει Μαριάν Ραχόη, αλλά ψηφίζοντας το Παρτίδο Ποπουλάρ ε, θέλει να γίνει Πρωθυπουργό ο Μαριάν Ραχόη. Το ίδιο ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι εκλέγεται και η καγκελάριος Μέρκελ. Αυτή είναι μια καινοτομία της ενδείξης της Σαββόνας που δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί γιατί ε, η συνθήκη ετέθησε ισχύ μετά τις τελευταίες ευρωεκλογέ, ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία από τους ε, Ευρωπαίους πολίτες την ώρα που θα ψηφίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε σήμερα αν είχαν διαβάσει τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα είχαν διαπιστώσει ότι απαντά σε πολλές ανησυχίες. Ταυτόχρονα ακούω διάφορες φωνές που λέγουν άμα είναι πολύ δύσκολο αυτά να εργαζόμαστε σε επίπεδο 27, υπάρχουν θέματα που είναι εχθρικά συστηματικά τα κράτη, πώς θα... Μα υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία. Έχουμε ήδη ε, προσφύγει σε αυτή για θέματα δευτερεύοντα, ας πάμε και σε άλλα θέματα. Ή αν μη τι άλλο, πριν αρχίσουμε να λέμε νέες συνθήκες, ας εφαρμόσουμε πλήρως την ισχύουσα. Και διαπιστώνω ότι σε θέματα που έχουν ενισχυθεί οι αρμοδιότητες της Ένωσης και που είναι κατεπίγουσα η κατάσταση και χρειαζόμαστε κοινέ πολιτικές, ε, παράδειγμα στην ενέργεια, στη μετανάστευση, στην εξωτερική, ε, στην ΚΕΠΑ και στην ΕΠΑΑ. Πού ροπέχουμε ακόμα από το να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις νέες δυνατότητες που μας επιτρέπει η συνθήκη. Η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης είναι κατακαιρματισμένη, θρύψαλα η πολιτική αμήνης δεν έχει κάνει ούτε σπιθαμή προόδου. Ενώ στη συνθήκη της Λισαβόνα έχουμε βάλει διατάξεις πάρα πολύ ευέλικτες, ε, ρεαλιστικές, με διάφορα βάρβαρα ονόματα, ξέρω εγώ, ε, μόνιμες επιτροπές κτλ. Αλλά μπορούν τα κράτη-μέλη, αν θέλουν, να προχωρήσουν περισσότερο, να τις αξιοποιήσουν. Αν θέλουμε λοιπόν, πώς να το πω τώρα, να προβληματιστούμε σοβαρά και να αρχίσουμε ε, πολιτική πρωτοβουλία για σύνταξη νέας συνθήκης, θα πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά τι, προβληματική, τι πρόβλημα μπορεί να σημαίνει μια νέα ευρωπαϊκή συνθήκη. Εντάξει, μια πολυτεχνική συνθήκη πάντα είναι δυνατή. Παρένθεση. Η συμφωνία της 21ης Ιουλίου που ανέφερα προηγουμένως, ανεξάρτητα από το όνομα, το νομικό, ήταν συνθήκη. Γιατί χρειάστηκε να κυρωθεί από κοινοβούλια. Κλείνει η παρένθεση. Ένα ερωτηματικό τώρα, εν παρόδο. Ποιος ημών γνωρίζει τι έγινε με την κύρωση της μήνης συνθήκης που είχε εγκριθεί πέρσι το, ε, φέτος το, το, την Άνοιξη. Έκθεση Μπροκ Φερχόφστατ, ξέρετε συνάδελφοι. Δεν θυμάμαι το άρθρο της συνθήκης, ε, αλλά ήταν για να αλλάξει η διατύπωση της διάταξης που απαγορεύει τη διάσωση, το bailout. 136, μάλιστα. Τι έγινε με την επικύρωση αυτού, ρώτησα προχθές και μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία χώρα που να έχει αρχίσει αυτή την επικύρωση της μικροσυνθήκης, που είναι τρεις γραμμές, έτσι στοιχηματίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε τις 27 κυρώσεις. Γιατί είμαι πεπισμένο ότι με τις 27 για κανένα θέμα δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουμε. Ούτε καν, πούμε, για την είσοδο της Κροατίας. Δεν πρόκειται ποτέ. Γιατί υπάρχει πάντα κίνδυνο σε κάποια χώρα μέλος να υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα που τσακώνεται η ε, συμπολίτευση με την αντιπολίτευση και δεν μπορούν να τα βρουν στο κοινοβούλιο ή στο δημοψήφισμα γιατί ξέρω εγώ είναι αγανακτισμένοι, έρχονται και αγανακτούν και δεν απαντούν στο ερώτημα του δημοψηφίσματος. Όλα αυτά τι σημαίνουν. Αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια πρωτοβουλία σημαντικής αναθεώρησης της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε από το να τολμούμε να ε, προβληματιζόμαστε και να θέτουμε σημαντικά ερωτήματα. Τρία για να μην μακρηγορήσω. Πρώτον, εκείνοι που προτείνουν τροποποίηση της συνθήκης είναι πρόθυμοι να προτείνουν ε, την εγκατάλειψη της ομοφωνίας για την κύρωση της νέας συνθήκης. Αν όχι, χαμένος κόπος, δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Αν είναι πρόθυμοι να απεμπολίσουν την ομοφωνία, σημαίνει ότι είναι πρόθυμοι να απεμπολίσουν το ίδιο το δικαίωμα βέτο. Προφανώς. Ο καθένας βέβαια είναι πρόθυμος να το ζητήσει από το διπλανό του, αλλά εντάξει. Δεύτερη ερώτηση. Ε. Είναι πρόθυμοι να υλοποιήσουν σημαντική συνθήκη που θα χώριζε την Ευρώπη στα δύο. Θα τη δίχαζε και με ποια κριτήρια, πέρα από κάποια δευτερεύοντα. Είναι δύο συζητήσεις που πρέπει να γίνουν και πάντα τις αποφεύγουμε. Ε, κάποιες νήξεις κάνουμε, αλλά επί της ουσίας δεν κάνουμε συζήτηση. Δύο Ευρώπες θέλουμε η μία. Ποια είναι η χρήσιμη Ευρώπη εντό εισαγωγικών, εκείνη του ευρώ ή των 27 των χωρών που έχουν καλή διαχείριση που είναι μερικά στο ευρώ και μερικά όχι κράτη, οι χωρε που έχουν κακή διαχείριση, γιατί είναι και αυτε χωρε ευρωζώνη και καποιε αλλε που δεν είναι. Ή μήπω η Ευρώπη που θέλουν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο των Ευρωπαϊστών, η Συμμαχία των Προθήμων που λένε και οι Αμερικανοί φίλοι μα ή η Ευρώπη των Ευρωχλιαρών. Ποια είναι η καλή Ευρώπη και η χρήσιμη και ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία για να έχουμε δύο κύκλους. Πρώτη εθνική, δεύτερη εθνική. Και κάτι ακόμα. Γιατί ακούω για την ομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρσρούης, που είναι πολύ σημαντική και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Όπως και όλα τα συνταγματικά δικαστήρια κατά τα άλλα των υπολείπων 26 κρατών. Είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες έχουν ισχύ ευρωπαϊκού συντάγματος, ακόμα και αν δεν λέγονται έτσι, και θα κυριαρχούν συστηματικά επί των εθνικών συνταγμάτων. Εάν είναι καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματα, ίσως να μπορέσουμε να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Αν όμως δεν έχουμε απαντήσει, δεν έχουμε συζητήσει αυτά τα τρία, προσοχή και να μην ανοίγουμε τέτοιες ιστορίες. Τελειώνω. Λέγοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε μήπως έχει έρθει η ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να αποφανθεί σε αυτή τη συζήτηση η οποία αρχίζει και έχει και θετικά στοιχεία. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι γίνεται σε σαφρά θεμέλια, με κακή κατάσταση της σημερινής κατάστασης, και αφήνουν να εννοηθεί, να ελπίσουμε ότι η σημερινή οικονομική κρίση μπορεί να έχει θεσμική επίλυση, ενώ κάθε θεσμική λύση θα χρειάζεται πέντε χρόνια, για να μην πω δέκα. Οπότε χρειάζεται ξανά ένταξη αυτό το θέμα σε μια πιο ρεαλιστική προοπτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαμασούρ. Ήταν μια πραγματικά έξοχη ε, εισήγηση και πιστεύω ότι πρέπει σε βάθος να σκεφτούμε όχι μόνο σήμερα στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης αλλά και ιστερότερα αυτά τα θέματα. Νομίζω τα ουσιοδέστερα θέματα αναφέρατε και έτσι πρέπει έτσι να τα δούμε και πρέπει να τα σκεφτούμε σε βάθος. Υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις. Ο κύριος Κουαλτιέρη πρώτος, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λαμασούρα από πλευράς μου τον ευχαριστώ διτά για την εργασία του και το έργο του για αυτό το έγγραφο εργασίας έγκαιρα υποβάλλεται και είναι πολύ ουσιώδη τα σχόλια. Δεν θα αντιδράσω σε όλα τα σχόλια του τώρα. Ήδη έχει γίνει πολλά και σε αυτό στο παρελθόν και χαίρομαι που αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή κατανόησε επιτέλους την ανάγκη που υφίσταται να ανταποκριθούμε σε αυτά τα οποία προτείνει ο κύριος Λαμασούρ και πρέπει να τοποθετηθούμε και να αναφέρουμε ποιες είναι οι απόψεις μας για αυτά τα θέματα και τι μπορεί να γίνει με τις συνθήκες Λισαβόνας. Πολλά μπορούν να γίνουν με τις συνθήκες Λισαβόνας. Και θα ε, απαιτηθούν και πολλά για μια τροποποίηση της συνθήκης. Δεν θα τοποθετηθώ επ' Αυτή η συζήτηση αντανακλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και σε σχέση με την πράσινη βίβλο και που θα ληφθούν υπόψη και αύριο και στο εγγύς μέλλον. Και για τα ευρωομόλογα και για την, ε, τις αναγκαίες αλλαγές συνθήκης δεν, δεν λέει η Επιτροπή αν τελεσίδικα θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση συνθήκη ή όχι. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είναι εκείνη που πρέπει να τοποθετηθεί επ' αυτόν. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, υπερβολικά σημαντικό για να συζητηθεί εδώ και τώρα μόνο. Και θα ήθελα να επικεντρωθώ στο έγγραφο εργασία του κυρίου Λαμασούρ και να πω κάποια πράγματα. Υπάρχει μια αντίφαση που αντανακλάται σε αυτό το έγγραφο εργασίας υφίσταται και μια αντίθεση αμφισημία στη συνθήκη και όσον αφορά και τι εξουσίε του Κοινοβουλίου και λόγω τη συνθήκη τη Λισαβόνα ταυτόχρονα όμω έχουμε και το νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω δημιουργεί μια ασύμετρη σχέση μια μεταβλητή γεωμετρία μεταθέτει το κοινοβούλιο από το επίκεντρο του κύκλου αυτής της ε, συζήτησης και το μεταθέτει εκτός ε, επικέντρου. Και αυτό δημιουργεί την ασύμετρη σχέση πραγμάτων. Υπάρχει μια αντίφαση σε σχέση με το άρθρο 10 και την εκπροσώπηση των πολιτών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούνται από τους ερετούς εκπροσώπους στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Ευρωκοινοβουλίου και μέσω αυτής της άσκησης εξουσιών έχει επίσης το Ευρωκοινοβούλιο νομοθετικά δικαιώματα για κάποιες πολιτικές, για κάποιους τομείς πολιτικών που δεν συμπίπτουν υποχρεωτικά και δεν υπάρχει επικάλυψη. Πώς ασκεί λοιπόν το ρόλο της ω ερετό εκπρόσωπος ε, των ε, πολιτών τη Ευρώπη στο Ευρωκοινοβούλιο και για αποφάσεις που δεν υφίστανται στη, ε, στην κανονική νομοθετική διαδικασία. Πώς μπορούμε να πληρώσουμε, να, να καλύψουμε αυτό το κενό. Υπάρχει εδώ θέμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί και πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό. Έγκαιρα λοιπόν και σε πολύ καλή χρονική στιγμή υποβάλλεται το έγγραφο του κυρίου Λαμασού για να δούμε πώ μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό. Πρώτον λοιπόν, δεν θεωρώ, δεν πιστεύω ότι αυτή η τάση που υφίσταται προς ε, μια κοινοτική μέθοδο, δηλαδή εφόσον η Ένωση θα αντιμετωπίζει νέα θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από την παραδοσιακή διαδικασία και θα πρέπει να ληφθούν διαφορετικές μέθοδοι υπόψη. Για παράδειγμα, η διακυβερνητική διάσκεψη που θέτει όμως τους πολίτες εκτός. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συντονίσουν, λέει, την ε, οικονομική τους πολιτική μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όμως τι γίνεται εκτός αυτού του πλαισίου. Δεν θα πρέπει εκτός αυτού του πλαισίου να γίνονται αυτά. Προβλέπεται λοιπόν η διακυβερνητική, το διακυβερνητικό επίπεδο. Ανοίγει λοιπόν η συζήτηση εδώ για να δούμε τι μπορεί να γίνει ώστε να επανέλθει αυτό το ζήτημα στο κοινοτικό πλαίσιο, στις κοινοτικέ αρμοδιότητες και να υπάρξουν κοινοτικές ε, ε, ενωσιακές ε, πρωτοβουλίες και πολιτικές. Θα πρέπει να δομηθεί ένας διάλογος και με τα άλλα όργανα τα οποία θα είναι αρμόδια προς λήψη απόφαση. Δεν είναι λοιπόν θέματα τα οποία περιορίζονται και για το ότι το 15 ή 16 δεν συνάδουν ή δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά. Όπως είπε ο κύριος Λαμαζού υπάρχει τεχνική υφή ε, έλλειψη ή κενό για την υλοποίηση την εφαρμογή άρθρων της συνθήκης και πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα έπρεπε να υποβάλει προτάσει προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έπρεπε να δημιουργήσει, να δομήσει ένα διάλογο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό προτείνεται ε, στην έκθεση που εγώ έχω την τιμή να συντέξω όσον αφορά τι πολιτικέ αυτέ και μετά την συνθήκη τη Λισαβόνας. Όταν κάνουμε λόγο για ένα τέτοιο είδου στρατηγικό διάλογο δεν μπορεί να είναι μόνο υπό το πλαίσιο του άρθρου 36 που αφορά διάλογο του Κοινοβουλίου με το ε, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Όχι, πρέπει να ξεκινήσουμε έναν διάλογο που δεν ε, ε, αποκλείεται από τις συνθήκες ούτε καλύπτεται αυτή τη στιγμή. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικής μορφής διαλόγου από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει, αντανακλώντα τι ευαισθησίε του Ευρωκοινοβουλίου έναντι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να βρούμε, να εξευρεθεί ο πιο σωστό διάλογο που πρέπει να δομηθεί. Και μετά η Σύνοδο τη Ευρωζώνη. Εδώ ένα ε, τεχνική υφή σχόλιο. Ίσως ο κύριο Λαμασούρ ήταν υπερβολικά γενναιόδωρο εντό εισαγωγικών, διότι κάνει λόγο και αναφέρει ότι εφόσον θα έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα έχουν εγκριθεί κάποια συμπεράσματα από αυτό το ε, θεσμικό όργανο πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Τα θεσμικά όργανα πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση τις συνθήκες τις ίδιες. Από νομική πλευράς λοιπόν η Σύνοδος της Ευρωζώνης δεν είναι ένα θεσμικό όργανο. Είναι ένα ας το πω έτσι ξεχωριστός θεσμός που λειτουργεί, που δεν έχει μορφή θεσμικού οργάνου, διότι δεν βρίσκεται ε, μορφή συνθήκης η εντολή και δεν προβλέπεται από μια συνθήκη η εντολή που έχει. Τούτου λεχθέντος δεν, δεν σημαίνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να αρνηθεί την ύπαρξη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης. Όχι, είναι ένα γεγονός, υφίσταται αυτό και, αυτό και πρέπει να έχουμε και διάλογο που θα δομήσουμε με αυτό. Όμως ε, πρέπει να δούμε το παράδοξο το οποίο υφίσταται εδώ, διότι κάποιοι θέλουν να αλλάξει η συνθήκη ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούν ήδη τώρα σήμερα να γίνουν. Και η μόνη απόφαση που ελήφθη σε σχέση με τη Σύνοδο του Οκτωβρίου ήταν να δημιουργηθεί η ως όργανο αυτή η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ε, και μάλιστα αναφορά σε μια αμελλοντική τροποποίηση της ε, συνθήκης. Σε αυτή την ασυμμετρία αναφέρομαι όσον αφορά τις σχέσεις ε, με το όργανο που εκπροσωπεί τα 17 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης σε σχέση με τα υπόλοιπα. Θα πρέπει εδώ να δούμε πώς μπορεί το Ευρωκοινοβούλιο να διαδραματίσει ένα ξεχωριστό ρόλο όταν αφορώνται θέματα τα οποία αναφέρονται στα 17 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Αν διαβάσετε το άρθρο που προβλέπει την ε, λήψη απόφασης από πλευράς του Συμβουλίου για τα 17 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Μία από τις αναφορές ε, είναι η κανονική νομική διαδικασία βάσει της συνθήκης που ρητά προβλέπει μια κανονική διαδικασία με το Συμβούλιο συμπεριλαμβάνοντας ε, ψήφιση από 17 κράτη-μέλη ενώ οι ψηφοφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τα 27 κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επ' αυτών των θεμάτων πρέπει να πω ότι εργάστηκα ε, και συνέταξα μια έκθεση για το αντίστοιχο άρθρο. Θέλουμε να δούμε το άρθρο αυτό και πώς μπορούμε να συμμορφωθούμε. Ήδη πρέπει να ε, πούμε ότι όταν έχουμε θέματα διορισμών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όταν ε, συμπεριλαμβάνεται η απόφαση των 17 κρατών που εκπροσωπούνται στην ε, ε, νομισματική ένωση, στην Ευρωζώνη, ενώ έχουμε 27 κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στο ενωσιακό επίπεδο, πρέπει να δούμε τι γίνεται εναντί των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα 17 κράτη-μέλη και κατά συμμετρική αντιστοιχεία τι γίνεται σε σχέση με αποφάσεις που λαμβάνονται από τα 27 κράτη-μέλη. Πρέπει να διασφαλιστεί μια ισόρροπη σχέση η συμμετρία και πρέπει αυτά να δούμε και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τα θέματα που καλύπτονται ακριβώς από την έκθεση Λαμασού. Είναι θέματα που εκκρεμούν και δεν έχουν επιληθεί. Ο ρόλος ε, της ΥΠΑ ε, της εκπροσώπου ή του ΥΠΑ του εκπροσώπου στις ε, συζητήσεις στην Ολομέλεια. καμιά φορά υπάρχει και παρακολούθηση, συνοδεύεται και από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. δεν πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην παραδοσιακή ε, οδό και ευθεία όταν έχουμε την ύπατη, ε, ε, ύπατο εκπρόσωπο κυρία Άστον. Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι διεργασίες και οι διαδικασίες έναντι αυτών των δύο αρμοδιοτήτων που έχει ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ως ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί των άλλων θεμάτων δεν θα τοποθετηθώ. Πρέπει να έχουμε την ευκαιρία ω Κοινοβουλευτική Επιτροπή να συζητήσουμε αυτά τα θέματα σε μεγαλύτερο βάσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχω πιστεί και με, έχει, με πείθει αυτό ότι πρέπει να αναβάλουμε τα θέματα προ συζήτηση μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μα. Και για τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν πριν από την ψήφιση προ έγκριση. Ε, εγώ είμαι εισηγητή για το ένα, ο άλλο ο άλλος είναι ο κύριο Ντάφ σε σχέση με τι αλλαγέ ε, διαδικασία διαδικαστικά των κανόνων και κανονισμών. Πρέπει να αναβάλουμε λοιπόν ώστε να διεξαχθεί σε μεγαλύτερο βάσος, βάθος όπως ε, θα συνείδε αυτή η συζήτηση. Και έτσι λοιπόν ήδη ε, συμφωνούμε με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ότι θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση μαζί τους στις 11.30 για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε κάποια σχόλια τώρα, σύντομα σχόλια όμως, ε, θεμάτων που μας αφορούν. Δεν θα πρέπει να μακρηγορούμε. Ο κύριος Ρανζέλ πρώτος. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι θα μιλήσω στα πορτογαλικά, μια και έχουμε πολλούς πορτογαλόφωνους. Θα είμαι πολύ σύντομος, ευθυγραμμιζόμενος και στις παρατηρήσεις του κυρίου Λαμασούρ. Θα ήθελα να επισήσω την προσοχή σε ένα σημείο. Εγώ θεωρώ ότι αξίζει εδώ να λάβουμε υπόψη τις, ε, τα θέματα έναντι του Συμβουλίου. Διότι παρότι για μας είναι πολύ σημαντικό το Συμβούλιο να μας δίνει πληροφορίες και να μας ενημερώνει, για την παρουσία του ίδιου του ε, Προέδρου του Συμβουλίου και από την άλλη πλευρά, από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου, για να υπάρξουν επεξηγήσει για τι συνόδου κορυφή και για τη σύνοδο του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εμεί θεωρούμε ότι το Συμβούλιο είναι ένα υπεύθυνο όργανο που πρέπει να λογοδοτεί έναντι του Κοινοβουλίου. Δεν γίνεται όμω ε, πάντα αυτό. Δεν είναι υπεύθυνο και δεν λογοδοτεί πάντα το Συμβούλιο στο έναντι του Κοινοβουλίου. Είναι ισότιμο όργανο on equal footing όπω αναφέρω αναφέρεται νομοθετικά έναντι του Κοινοβουλίου. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το συσχετισμό μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου. Γιατί καμιά φορά δίνει την εντύπωση ότι εξαρτάται το Συμβούλιο από το Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ δύο συνιστώσεις πρέπει να δούμε έναν του Συμβουλίου. Το εκτελεστικό επίπεδο και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και σε σχέση με τις, ε, την πολιτική, ας το πω έτσι, ηγεσία που ασκείται από το ε, Συμβούλιο, έτσι να υπάρξουν κάποιες ε, επεξηγήσεις έναντι του ε, Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αν δεν συμβαίνει αυτό, θα τεθεί το Συμβούλιο σε μια θέση όπου δεν θα υπάρχει ισότιμη σχέση Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και γι' αυτό θα πρέπει αυτή η παρατήρηση να ληφθεί υπόψη σε σχέση με την έκθεση ή στο σχέδιο έκθεσης που υποβάλλεται από τον κύριο Λαμασούρ. Δεύτερη πτυχή που θεωρώ ότι εδώ είναι πολύ σημαντική είναι η σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Εδώ θα πρέπει να πω ότι είναι φυσικό το Συμβούλιο να έχει άμεση σχέση και συσχετισμό με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Διότι αυτό το οποίο, αυτό, εκείνος ο οποίος ελέγχει τη στάση των μελών του Συμβουλίου, τη στάση και τις συμπεριφορές των ε, μελών του Συμβουλίου είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια που ε, εκπροσωπούν, εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις τους. Δεν είναι λοιπόν το Συμβούλιο το οποίο έχει μόνο την συνιστόσα του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και τη συνιστόσα των Εθνικών Κοινοβουλίων έτσι υπό τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας πρέπει να δούμε την ισότιμη σχέση equal footing μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι όμως ε, ε, θέση απλά λογοδότησης ή ευθύνης. Και γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι καμιά φορά είναι διστακτικό ή επιφυλακτικό να ε, δώσει, ε, να υπάρξει άμεση αντίδραση από το Συμβούλιο σε ερωτήσεις εναντί του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως για παράδειγμα μια γερουσία ή εναντί ενός κοινοβουλίου. Αν είναι δυνατόν με ένα νομοθετικό θέμα, σώμα το οποίο θα ήταν ισότιμο απέναντι του Συμβουλίου θα έπρεπε να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει γίνει. Υπάρχει αυτή η αμφισημία. Αυτή η αμφισημία ε, που ε, υφίσταται. Το Συμβούλιο είναι ένα ε, όργανο το οποίο δίνει πολιτικές κατευθύνσεις και κατευθύνει την πολιτική. Εδώ τουλάχιστον στο επίπεδο το κυβερνητικό. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν κάποια πράγματα έναντι του Ευρωκοινοβουλίου να α, επεξηγούνται. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, να δούμε αυτή τη συνιστόσα του, του συσχετισμού μεταξύ του Συμβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, να εμβαθύνουμε σε αυτό το συσχετισμό, σε αυτή τη σχέση, διότι είναι ακριβώς αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων έναντι των εθνικών κυβερνήσεων να δίνεται η εντολή και μετά να ασκείται ε, έλεγχος ώστε να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις έναντι των κοινοβουλίων για αυτά που κάνουν. Στο ίδιο επίπεδο πρέπει να δούμε τις δράσεις του Συμβουλίου έναντι αυτών των ε, εθνικών κοινοβουλίων. Και απέναντι στο Ευρωκοινοβούλιο, να δούμε τις αρμοδιότητες που υπάρχουν, πώς μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε. Εδώ, στην ίδια την έκθεση, δεν είναι μόνο θέμα της έκθεσης, αλλά είναι και το θέμα της, του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα μπορέσουν οι συνθήκες να προσαρμοστούν και με ποιο τρόπο. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να βάλουμε τα πράγματα το κάθε ένα στη σωστή του θέση. Εμείς δεν πρέπει να, αποκλίνουμε, να αποκλείσουμε κάποιες τεχνικές τροποποιήσεις ή προσαρμογές, ιδιαίτερα όσον αφορά το πρωτόκολλο 14 για αυτές τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες. Άλλο θέμα εν κατακλείδη είναι το εξής το Κοινοβούλιο σε σχέση με την εξέταση των θεμάτων του, της ζώνης ευρώ. Δεν συμφωνώ με τον, τον ορισμό του συναδέφου Γκουαλτιέρη για μια ιδιωτικού χαρακτήρα ή ξεχωριστού χαρακτήρα λέσχη ή όργανο. Με βάση τις συνθήκες όλα τα κράτη και τα 27 κράτη-μέλη εδώ πρέπει να δούμε ότι πρέπει να ε, έχουν την αρμοδιότητα έναντι των θεμάτων ε, ευρώ. Δεν μπορούμε να θεσμοθετήσουμε ξεχωριστά ε, κάποια πράγματα σε ένα στεγανό ε, της ε, Ευρωζώνης συμπεριλαμβάνοντας ε, τις χώρες που έχουν και opt-out αυτοεξαίρεση όπως τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο πώς θα αντιμετωπίσουμε τους συναδέλφους των χωρών που δεν βρίσκονται στο ευρώ ή εκείνες τις χώρες τους συναδέλφους από εκείνες τις χώρες που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο ευρώ αυτά τα θέματα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν αλλά θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτά για μια μελλοντική ευκαιρία όταν θα έχουμε περισσότερο περισσότερο χρόνο να εμβαθύνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Σδάφ. Um, well... Λοιπόν, βεβαίως ευγνωμονούμε τον Αλέ Λαμασούρ για την τόσο εύστοχη και εχμηρή έκθεσή του. Πάντα μας εμπνέουν τα όσα λέγει. Νομίζω έχει αποκλίνει από τη έκθεση έτσι, με τη στενή έννοια. δεν πειράζει αυτό, καλό είναι. Αν βρισκόμαστε στα πρόθυρα συντακτική συνέλευση θα πρέπει το Κοινοβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε το εύρος ε, της συμφωνίας που θα προκύψει από τη συντακτική συνέλευση να είναι αρκετά μεγάλο έτσι ώστε να διευκολύνει την εξέβριση ε, συνένεσης. θα πρέπει να υπάρχει η ευκαιρία και να δράξουμε την ευκαιρία ε, διόρθωσης κάποιων σφαλμάτων που κάναμε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί έχουμε διαπιστώσει και αναγνωρίσει ότι υπάρχουν και στρεβλά. Αλλά υπάρχουν και παραλήψεις και χρειάζεται ίσως και συμπλήρωση να μπουν κάποια πράγματα που δεν λέει η συνθήκη. Αν ήταν χτες εδώ παρόν ο κύριος Λαμασούρ που συζητήσαμε το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και την Τσεχία για τη συνθήκη της Λισαβόνας θα του άρεσε η συζήτηση ε, για την ανάγκη να αλλάξουν οι διατάξεις για τη θέση σε ισχύ οποιασδήποτε μελλοντική συνθήκη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ε, και θα χρειαστεί να επανέλθουμε σε αυτό. Ένα δεύτερο που θεωρώ εξαιρετική ιδέα και είχε συμφωνηθεί στη συντακτική συνέλευση του το Ζισκάρ είναι να διαχωριστεί, να σπάσει το Συμβούλιο Υπουργών να ε, υπάρχει και ε, ένα νομοθετικό σώμα, ας πούμε, και ένα εκτελεστικό σώμα στο Συμβούλιο. Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ε, αμήνης ή σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης, όπου το Συμβούλιο έχει συντρέχουσες εκτελεστικές εξουσίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι σχέσεις του με το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετικής ποιότητας από τις σχέσεις που έχουμε τώρα εμείς με το Συμβούλιο. Όταν ως νομοθέτης. Καλή ιδέα λοιπόν αυτή και θα πρέπει να επανέλθουμε. Επίσης πιστεύω ότι η ιδέα δύο σωμάτων, δύο πρόεδρων μάλλον, ε, ο μόνιμος λεγόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν μάλλον σφάλμα. Και τότε εγώ το είχα υποστηρίξει, αλλά έχω αλλάξει γνώμη εκ τότε. Όχι λόγω του προσώπου του κύριου Βαν Ρομπέι, τον οποίο θαυμάζω και σέβομαι και τιμώ, αλλά εν μέρη επειδή είναι οικονομολόγος ο ίδιος και έχει αναμειχθεί στην οικονομική κρίση με τρόπο ο οποίος δεν προβλέπεται από τη συνθήκη και ήρθε να υποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό και μάλιστα σε κάποιο ανησυχητικό βαθμό το ρόλο που του αναλογεί και έχει υποκαταστήσει περίπου τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ρόλο του στην προσπάθεια ε, επίτευξης ε, δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάκαμψης. Αυτό το είδα και στα θέματα των εξωτερικών υποθέσεων, όπου και ο Μπαρόσο και ο Φαν Ρομπέι ε, διαγωνίζονται ή ε, ανταγωνίζονται για τις ίδιες επιτροπές για να προεδρεύσουν και οι δύο. Και είναι πρόβλημα αυτό. Και αν λένε ακριβώς το ίδιο θέμα και έχουν την ίδια θέση, ε, τότε τίθεται το ερώτημα γιατί να έχουμε δύο πρόσωπα σε αυτές τις θέσεις. Το πιο λογικό θα ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υποπτεύομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί το 2014 έτσι και αλλιώς. Αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε γι' αυτό σε συντακτική συνέλευση, δεν είναι του παρόντος, και να προετοιμαστούμε αναλόγως και κατάλληλα. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, Νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να αναγκάσουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να λογοδοτεί, να αναφέρεται στην Ολομέλεια. Και όχι σε μια διευρυμένη διάσκεψη των Προέδρων, που δεν είναι το σωστό όργανο, ούτε το σωστό και το κατάλληλο βήμα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα εθνικά κοινοβούλια, Υπάρχει κάτι που με ενοχλεί. Απλώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων για θέματα ευαίσθητα. Μα τι γίνεται με τη διάκριση των εξουσιών. Ε, νομίζω ότι εδώ υπέρχεται μια ε, σύγχυση και μια συσκότηση των αρμοδιοτήτων. Ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχω και άλλα σχόλια. Ε, συμφωνώ απολύτως ε, για το παράλογο του προγράμματος που αποφάσισε η Τσεντεού στη λειψία της προάλλες για την άμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πορείας άξιων πώς έτσι, ένα ε, υπεύθυνο πολιτικό κόμμα έδειξε τέτοια έλλειψη νυφαλιότητας. Εν πάση περιπτώσει. Καθώς φτάνουμε στο κατόφλι της συνέλευσης, όλα αυτά θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Ευχαριστώ. Grazie, Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε μια συζήτηση η οποία είναι λίγο πιο ευρεία από ότι τουλάχιστον το έγγραφο το οποίο βρίσκεται στη βάση. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις συνέπειες της υπάρχουσας συνθήκης και πριν καταφέσουμε νέες ιδέες καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι εκμετάλλευση γίνεται των υπαρχουσών προτάσεων που περιλαμβάνονται στη συνθήκη ιδιαίτερα στην περίπτωση ακριβώς των χωρών οι οποίες έχουν διάθεση να προχωρήσουν σε περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πράγματι έχουμε εφεύρει βέβαια εδώ και λίγα χρόνια την ενισχυμένη συνεργασία και τους τρόπους με τους οποίους η ενισχυμένη συνεργασία μπορεί να διεξαχθεί, να εξελιχθεί στα πλαίσια της συνθήκης. Σχετικά επίσης με το θέμα των αλλαγών της συνθήκης, με την ειδική πλειοψηφία, θα δούμε ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο είχε προκαλέσει, αν ενθυμίστε, ιδιαίτερα προβλήματα και κατά τη διάρκεια της τελευταίας συντακτικής συνέλευσης. Πάντως, η συζήτηση η οποία θα γίνει, έχω την αίσθηση ότι είναι σημαντική και παρουσιάζει προβλήματα και είναι μια συζήτηση η οποία θα ξεπεράσει σε σημασία αν θέλετε και σε ενδιαφέρον τη συζήτηση που γίνεται και που απασχολεί τους πολίτες σήμερα γύρω από την οικονομική περαιτέρω διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν διαφορές οι οποίες εκφράζονται στα πλαίσια των ρητορικών και από τις δύο πλευρές σε σχέση με τις νέες προτάσεις για τη συνθήκη σχετικά με την εθνική κυριαρχία και όλα αυτά ε, και διαρωτώ με αν ένα θέμα το οποίο θα βάζαμε εμείς προς συζήτηση με αυτούς τους όρους θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα. Εν πολλής τα γεγονότα μας έχουν προλάβει. Ενθυμίστε λίγο τα επιχειρήματα τα οποία είχαμε ακούσει την εποχή της συνέλευσης ότι δεν θα πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις με τον πρόεδρο του Συμβουλίου διότι θα του αποδώσει περισσότερη αν θέλετε ε, αντιπροσωπευτικότητα αυτό δεν είναι σωστό. Έχουμε κάποιες σχέσεις βέβαια, μορφές συγκεκριμένες σχέσεων με τον πρόεδρο του Συμβουλίου και άκουσα από τους συναδέλφους ότι η συζήτηση με την Προεδρία του Συμβουλίου έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί αποστέλει προς όλους τα σωστά μηνύματα ότι στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση το αγκυρώνουμε στην κοινοτική μέθοδο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. και γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν έχουν σχέση με αυτά τα οποία πιστεύει ο κόσμος ότι κάνουν τα κράτη-μέλη, δηλαδή σκοτεινές, υπόγειες διαπραγματεύσεις, κρυφίες διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στη φάση αυτή όπου ο Βαν Ρομπόι έχει διάθεση να συνεργαστεί. Σχετικά τώρα με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ιδιαίτερα αν δούμε τι κάνουμε στο κοινοβούλιο μας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την οικονομική διακυβέρνηση. Υπάρχει δυνατότητα να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε καλύτερα με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Και όπως είπαν οι συνάδελφοι, κάποια από τα μαθήματα της πολωνικής πρωτοβουλίας στο δημοσιονομικό επίπεδο θα είναι χρήσιμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετές αντιφατικές ιδέες σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση και για τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλέξουμε περισσότερο τα κοινοβούλια των κρατών μελών ε, και σύμφωνα πάντα με την διοργανική συμφωνία. Ε, υπό ποιους όρους θα μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με τα κοινοβούλια των κρατών μελών έτσι ώστε να μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε έτσι περαιτέρω ε, τις σχέσεις μας με τα κοινοβούλια. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα μαθήματα της πρωτοβουλίας της Πολωνικής για τον προϋπολογισμό, τα οποία δεν πήγαν καθόλου, θα έλεγα, η πρωτοβουλία μάλλον δεν πήγε καθόλου άσχημα και υπόσχεται αρκετά. Και ας δούμε τι θα γίνει και με την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις. Αν θέλουμε εμείς να ορίσουμε σωστά τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες αυτές, νομίζω ότι τότε θα έχουμε ξεπεράσει ένα πρώτο σκόπελο. Ευχαριστώ κύριε Φεσκόφσκι. Ο κύριος Γκουερέρο έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Δεν θα επιστρέψω στα θέματα ουσίας, διότι υπήρξαν πολύ αξιόλογες παρεμβάσεις ούτως ή άλλως, πέρα από την αξιολογότατη παρέμβαση του κυρίου Λαμασού. Υπήρξαν όμως τρεις ή τέσσερις ήδη παρεμβάσεις που ίσως εδώ πρέπει να δούμε ότι επικεντρώθηκαν κάπως στο θέμα του τι είναι αυτό το οποίο συζητάμε σε αυτή την έκθεση. Και επιτείνω συζητήσαμε ακριβώς σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Η έκθεση είναι για βελτιώσεις των θεσμικών σχέσεων σύμφωνα πάντα με τις συνθήκες της Λισαβόνας. Και ένα μέρος της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από ενδεχόμενες αναθεωρήσεις ε, μεταρρυθμίσεις της συνθήκης. Αυτονόητο είναι φυσικά ότι και τα δύο αυτά θέματα διανοητικά συνδέονται και αλληλοσυναρτώνται και στο πολιτικό επίπεδο. Καθώς όμως δεν είναι δυνατόν όλα τα μέλη που είναι σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή να έχουν τις πληροφορίες που θα δώσω, θεωρώ σκόπιμο να ενημερώσω τα μέλη αυτά σχετικά με αυτά τα θέματα. Όπως γνωρίζετε Πρόεδρε, εχθές, εχθές οι συντανιστές δώσαμε εντολή στον Πρόεδρο να έρθει σε επαφή με την Πρόεδρο της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΚΟΝ ώστε να προσπαθήσει να διοργανώσει μία συνεδρίαση με τους συντονιστές της ΕΚΟΝ και της ΑΦΚΟ ώστε να ξεκινήσει από κοινού αυτό το εγχείρημα μέσα στο πλαίσιο τουλάχιστον της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων μια διαρκής, ένας διαρκής προβληματισμός για τη διαδικασία αναθεώρησης των συνθήκων γύρω από μια έκθεση ευέλικτη ιδέα πρωτοβουλία που προτάθηκε από τη σοσιαλιστική ομάδα πριν από κάποιου μήνε και που προφανώ θα μπορούσε να περιστρέφεται γύρω από σήμερα το πρωί κάναμε λόγο για προσανατολισμούς Προσανατολισμούς λοιπόν για μια ενδεχόμενη μεταρρύθμιση της συνθήκης όσον αφορά την ε, χρηματοοικονομική, την οικονομική διακυβέρνηση. Θα ήθελα να πω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε με την έκθεση του κυρίου Λαμασούρ ίσως έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτή η ουσιώδης όμως συζήτηση είναι ε, πολύ θετική και σκόπιμη για τη συζήτηση για τους προσανατολισμούς για τους οποίους δόθηκε εντολή στον πρόεδρο να έρθει σε επαφή με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Λαμασούρ διότι η ευκαιρία της έκθεσής του που αφορά στον κανονισμό έθεσε ορισμένα ζητήματα τα οποία φαίνεται να μην λαμβάνουν υπόψη όσοι επιμένουν για αλλαγή της συνθήκης. Κύριε Πρόεδρε, η συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Ο κύριος Λαμασούρ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση που δημιούργησε τη Συνταγματική Συνθήκη και είδαμε πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα και βεβαίως γνωρίζουμε ότι για να αλλάξουν οι συνθήκες πρέπει να υπάρξει Ευρωπαϊκή Συνέλευση αλλά η θεωρία ορισμένων ότι θα ανοίξουμε τις συνθήκες μόνο για ορισμένα άρθρα για να κάνουμε αλλαγή απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Εάν ανοίξει θέμα τροποποίηση των συνθήκων με συνέλευση θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου Δηλαδή ο καθένας θα έρχεται με τα δικά του θέματα σε οποιοδήποτε σημείο ενώ η συνθήκη όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Λαμασούρ δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Και βεβαίως παρακολουθούμε το Συμβούλιο να έχει οικειοποιηθεί τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως παρακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην παίζει το ρόλο της. Το Συμβούλιο δηλαδή να ασκεί και νομοθετικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες να υπάρχει κομφούζιο σε σχέση με την Ευρωομάδα ε, και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κάτι που δεν είναι σωστό και να ανακύπτει μείζον θέμα με το πώς αυτά ελέγχονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Διότι κύριε Πρόεδρε αυτό που θα συναντήσουμε μπροστά μας είναι η επανάσταση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και εγώ τη βλέπω να έρχεται. Επομένως έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έχει υποκαταστήσει τους πάντες και τα πάντα, κάνει ό,τι θέλει, δεν εφαρμόζεται στην ουσία η συνθήκη και έρχονται μέλη του Συμβουλίου και μας λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε τη συνθήκη. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Λαμασούρ ότι αν δεν είναι αποφασισμένοι να κάνουν πολιτικό βήμα μπροστά, δηλαδή να απαρνηθούν το δικαίωμα του βέτο και πολλά άλλα δικαιώματα που έχουν, να προχωρήσουμε στην κοινοτική μέθοδο εργασίας. Δεν βρίσκω κανένα λόγο και έχω την αίσθηση ότι το Κοινοβούλιο μας πρέπει να αντιδράσει να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή της συνθήκης πριν εφαρμοστεί η προηγούμενη. Διότι αυτό θα, έχει καταστροφικές συνέπειες αν λάβουμε υπόψη μας ότι εν μέσω κρίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει στις 21 Ιουλίου μετά ξεαποφασίζει μετά ξανααποφασίζει, δηλαδή υπάρχει ένα κομφούζιο και μία σύγχυση κύριε Πρόεδρε. Είναι ολοφάνερο ότι το Συμβούλιο και αυτοί που προτείνουν και η γερμανική πλευρά κυρίως που προτείνει αλλαγή των συνθήκων δεν είναι καθόλου αποφασισμένοι να αποποιηθούν δικαιώματα. Τότε τι είδου αλλαγή στη συνθήκη θέλουν να κάνουν. Εγώ ε, προτείνω κύριε Πρόεδρε επειδή δεν έχω την αίσθηση ότι σκοπεύει το Συμβούλιο να προχωρήσει κοινοτικά να κάνει βήμα προς την πολιτική ενοποίηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιδράσει στην προσπάθεια αλλαγής των συνθήκων με βάση συγκεκριμένα συμφέροντα συγκεκριμένων πλευρών. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι σοβαρό λάθος. Ευχαριστώ κύριε. Λοιπόν, ένα θέμα θα διαλέξω στο κείμενο του κυρίου Λαμασού. Θα ήθελα να πω ότι θα κάνει εντύπωση, συμφωνώ με τις ανησυχίες του για αυτά που είχε ο Βαν Ρόμπαϊ τον Ιανουάριο του 2010. Είχε πει ο Βαν Ρόμπαϊ ότι είναι ο υπόλογος προς το Συμβούλιο και όχι προφανώς προς την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από τις συναντήσεις του Συμβουλίου. <clears throat> ίσως χρησιμοποιεί τη λέξη responsible όχι μόνο σαν υπεύθυνο, όχι μόνο σαν υπόλογο, αλλά και σαν εναλλάξιμος. Η θέση του βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει εύκολα από το Κοινοβούλιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι πραγματικά υπόλογος. αν η θέση του υπήρχε όταν επικυρώθηκε η συνθήκη και αν είχε ευθύνη απέναντι στο Κοινοβούλιο θα μπορούσε να, το, μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τα θέματα που συζητούσαμε χθε σαν παράδειγμα για τα θέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τσεχίας και της Πολωνίας σε σχέση με τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε σχέση με τις εγγυήσεις τις οποίες έδωσε το Συμβούλιο προς την Ιρλανδία ανάμεσα στα δύο δημοψηφίσματα που έγιναν στη χώρα αυτή και αν έχουν κάποια αξία οι διαβεβαιώσεις αυτές. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Χέφνερ είναι ο τελευταίος και μετά θα μας απαντήσει ο κύριος Λαμασούρ. Ο κύριος Χέφνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Αλένα Μασούρ ο οποίος πάντα είναι πάρα πολύ παραγωγικός, ε, παράγει σκέψη και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ, όχι μόνο για τη δραστηριότητά του, αλλά και γιατί είναι πρωτοπόρο, σκέφτεται μπροστά ε, από τις εξελίξεις, έχοντας πάντα στο μυαλό του τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου και πώς μπορούμε να τα υπερασπιστούμε σε μια ε, μεταβαλλόμενη αρχιτεκτονική, πώς θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη συμμετοχή και δημοκρατική κυριαρχία. Τώρα θα συμφωνήσω με τους περισσότερους που μίλησαν. Δεν θέλω να μπω στον πυρήνα των προτάσεων που κάνατε στο πρώτο τμήμα. Τώρα κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση αρχής περισσότερο. Δεν έχω να προσθέσω πολλά γιατί πολλά υπόθηκαν και με κάλυψαν. Το μόνο που έχω να πω και μου φαίνεται σημαντικό γιατί δεν έχει καλυφθεί αρκετά. Οι ερμηνείς μπορεί να διαφέρουν, αλλά εμείς βασιζόμαστε αποκλειστικά με βάση τα σημερινά κείμενα για το τι είναι δυνατό και τι δεν είναι. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε, έτσι ώστε οι πολίτες στην Ευρώπη, άνδρες και γυναίκες, να συμμετέχουν ε, και πιο ενεργά. Και το λέω και ορμόμενος από τη γερμανική πραγματικότητα. Και η συζήτηση που γίνεται στη Γερμανία, παρακαλώ, δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Δεν είναι θέμα της κυρίας Μέρκελ ή κάποιων κομμάτων ή κάποιων συνεδρίων των κομμάτων. Στη Γερμανία υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση, βαριά πίεση και ρωτούν όλα αυτά που κάνουμε, με ποια νομική βάση τα κάνουμε, οικονομική διακυβέρνηση και όλα τα άλλα που έχουμε αποφασίσει για το ESM, EFSF. Μήπως χρειάζεται να προβληματιστούμε περισσότερο για τις διαδικασίες και τα θεσμικά όργανα. Πρέπει να σας πω ότι εγώ συμφωνώ με την άποψη αυτή και με την ανησυχία που υπάρχει ότι μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αλλαγή τροποποίηση της συνθήκης. Εάν θέλουμε να το κάνουμε καθαρά, δηλαδή με αρκετή ε, δημοκρατική νομιμότητα, με σωστές διαδικασίες που να έχουν και να, να προκαλούν, να γεννούν και την αποδοχή του κόσμου στην Ευρώπη. Γιατί στο μέλλον θα μας χρειαστεί αυτή. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να υπάρχει αποδοχή του κόσμου και ε, αναπομακρύνεται από μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι μια συντακτική συνέλευση δεν απαραίτητο εμπόδιο ή τροχοπέδι. Το αντίθετο, μπορεί να είναι και γκάζι, όχι φρένο. Εάν το οργανώσουμε σωστά, μπορεί να αποτελέσει μια διοργάνωση που σε μια χρονική στιγμή που έχουμε ένα δραματικό κατακαιρματισμό στην ευρωπαϊκή συζήτηση, να συγκεντρώσει κάπου τη συζήτηση και να την οργανώσει. Και μπορεί ενδεχομένως να παράγει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Μπορεί τυπικά και επίσημα να ισχύει ακόμα η ομοφωνία, αλλά η συνέλευση είναι ένας χώρος, ένας τόπος και μια διαδικασία που αναγκάζει τους συμμετέχοντες να βρουν μια κοινή λύση, η οποία ε, υποβάλλεται ως σύνολο τελικά. Και ε, ε, είναι και ένας χώρος που γίνεται σωστός προβληματισμός, έτσι με την απαραίτητη ηρεμία και νυφαλαιότητα σε βάθος. Και αν γίνει αυτή η συνέλευση, παρακαλώ να μην είναι μόνο τεχνική για να δώσει την ευλογία της ε, ε, σε συνθήκες που είναι τετελεσμένες, ας πούμε, εκ των προτέρων. Να έχουμε αρκετό χρόνο να το συζητήσουμε, γιατί μια τέτοια διαδικασία ακριβώς δεν οδηγεί πάντα μόνο σε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά παράγει και νομιμότητα και αποδοχή τελικά. Και έτσι η ευρωπαϊκή δημοκρατία μπορεί να αναζωογονηθεί και η κοινή μας και η έννοια του συνυπάρχειν που είναι τόσο απαραίτητη. Ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση, ο κύριος Κόρμπετ, ένας παλαιός ε, εκλεκτός συνάδελφος, ο οποίος εργάζεται ε, στις υπηρεσίες του κυρίου Βάνρομπα, ζήτησε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Δεν θα σας καθυστερήσω ιδιαίτερα. Ήθελα απλά να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία συγκεκριμένα τα οποία ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και τα οποία θα ήθελα να διευκρινίσω εκ μέρους του Βαν Ρόμπαϊ. Καταρχάς, η στάση του Βαν Ρόμπαϊ απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ομιλία, ομιλίες οι οποίες έγιναν από αυτόν σχετικά με την υποχρέωσή του να αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το πνεύμα αυτών το, τα οποία είπε είναι ότι η μοναδική νομικά δεσμευτική θα έλεγα αποστολή του μετά ε, τη λήξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά το συμπληρώνει αυτό με ακόμα περισσότερες δραστηριότητες και είδατε ότι κάτι τέτοιο επαληθεύεται. Έχει πάει και στη διάσκεψη των Προέδρων, έχει συναντηθεί επανειλημμένα με Προέδρους Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, έχει δεχθεί να απαντήσει προφορικές ερωτήσεις, γραπτές συγγνώμη ερωτήσεις, έχει επανειλημμένα συναντηθεί με τον κύριο Μπούζεκ, τον Πρόεδρο Μπούζεκ, έχει επαφές με τις πολιτικές ομάδες κτλ. κτλ. Έχει αναλάβει επίσης την υποχρέωση να αναφέρεται στο Κοινοβούλιο και μετά από τις συναντήσεις κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης. Κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια συνάντηση, περίπου παράλληλα με το Συμβούλιο, αναφέρεται και θα αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. το θέμα της συμμετοχής στην διάσκεψη των Προέδρων και όχι στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το οποίο σαν απόφαση ανήκει σε εσά, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο το αποφάσισε αυτό και όχι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο χρόνος ο οποίος μερικές φορές μεσολαβεί ανάμεσα σε μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην επόμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να είναι μακρύς. Ε, πολλές φορές είναι δύο εβδομάδες, οπότε συμφωνήθηκε ο πρόεδρος Βαν Ρομπάι να αναφέρεται άμεσα τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα στο κοινοβούλιο σας, σε μια ειδική συνάντηση η οποία μπορεί να οργανωθεί. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της εντολής του, τέτοιες συναντήσεις χαρακτηρίστηκαν σαν ολομέλειες από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν μίνι ολομέλειες για δύο ώρες στην, στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο ήμιση τώρα της εντολής του αποφάσισε το Κοινοβούλιο να ονοματίσει τις συναντήσεις αυτές διασκέψεις προέδρων ανοιχτή προς όλα τα μέλη. Αυτό είναι θέμα ε, του Κοινοβουλίου για λόγους προφανώς ισορροπίας ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Αυτό ήταν απόφαση του Κοινοβουλίου και όχι απόφαση του κυρίου Βαν Ρόμπαϊ πρέπει να το σχολιάσω αυτό, γιατί έγιναν κάποια σχόλια ε, που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει μια κάποια παρανόηση γύρω από το θέμα αυτό. Ένα τελευταίο σημείο για το εάν θα πρέπει να συμμετέχει στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις συζητήσεις μετά της ε, συναντήσεις του Συμβουλίου και αυτό συζητήθηκε με το Κοινοβούλιο στην αρχή της περίοδου εντολής και με τον Πρόεδρο και με τη διάσκεψη των Προέδρων. Τότε στις συζητήσεις αυτές ε, είχε, θα έλεγα, θεωρηθεί σωστό ότι αν πρέπει να έρχεται πριν και μετά από τις συναντήσεις του Συμβουλίου που είναι έξι περίπου κατέτος, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχει σε 12 συζητήσεις κατέτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή κάθε μήνα περίπου. Και αυτό θεώρησαν ορισμένοι ότι ίσως ε, θα τον βαρεθεί το ίδιο το Κοινοβούλιο να τον βλέπει κάθε μήνα να κάνει μια τέτοια συνάντηση ε, κάθε Τετάρτη πρωί. Και γι' αυτό το ίδιο το Κοινοβούλιο είπαν ότι ας αφήσουμε το υπάρχον σύστημα όπου ο Προεδρεύων της εναλλακτικής προεδρίας ε, της, του Κανονικού Συμβουλίου παρουσιάζεται ε, και αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί σύμφωνα με τις συνθήκες ε, τα συμβούλια τα ευρωπαϊκά προπαρασκευάζονται από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων όπως ξέρετε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόρμπετ. Ο κύριος Λαμασούρ πλέον για να τελειώσει η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους, για τις προτάσεις τους. Να ευχαριστήσω φυσικά και τον Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Θα έπρεπε να το πω από πριν ότι σχετικά με τον πρόεδρο Φαν Ρόμπαϊ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του έδωσε την εντολή να κάνει προτάσεις προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ε, στα πλαίσια ε, της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι προτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν και τροποποίησης της συνθήκης. Σε πολύ λίγες μέρες ή εβδομάδες έστω θα έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα την άποψη Βαν Τώρα κάποιες ε, απαντήσεις στα σχόλια των συναδέλφων. Θεωρώ ότι το παράδειγμα το οποίο έθεσε ο Γκουαλτιέρη στον τομέα της ΚΕΠΑ, στα πλαίσια δηλαδή του συγκεκριμένου στρατηγικού διαλόγου που ξεκινά με το Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι κάτι το θετικό και ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος με το Συμβούλιο. Αναφέρθηκε στην περίπτωση και της Ευρωζώνης ο κύριος Γκουαλτιέρη λέγοντας ότι δεν είναι στη συνθήκη. Μα φυσικά και υπάρχουν ρυθμίσεις στη συνθήκη ειδικέ και εφαρμόσιμες στη ζώνη ευρώ. Και η συνάντηση κορυφής της ζώνη ευρώ, δεν ξέρω ποιο είναι τώρα το επίσημο όνομα αυτού του οργάνου, είναι μια συνάντηση η οποία προς στιγμή δεν έχει θα έλεγα νομική βάση αλλά είναι προφανές ότι η επόμενη συνθήκη θα της δώσει μια τέτοια βάση γιατί και το Συμβούλιο δούλευε για 20 χρόνια χωρίς καμία νομική βάση. Η Άγγελα Ράγγελ είπε και έχει ε, δίκιο ότι το Συμβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών δεν είναι υπόλογο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έννοια την οποία σημείωσε και ο συνάδελφος Μπρόνς που μας μίλησε για τις εναλλακτικές έννοιες της λέξης της αγγλικής responsible. Πράγματι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βρίσκονται σε διάλογο ε, σε νομοθετικό επίπεδο σαν δύο κοινοβουλευτικά σώματα, το Άνω και το Κάτω Κοινοβουλευτικό Σώμα. Και είναι απολύτως θεμητό η διαδικασία, σαν παράδειγμα, των επικαίρων θεμάτων, ε, την οποία έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην εφαρμόζεται με το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συνδιαλεγόμεθα με το Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι ένα νομοθετικό όργανο, δεν είναι υπόλογο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μία μορφή θα έλεγα συλλογικού εκτελεστικού οργάνου που λαμβάνει αποφάσεις λίγο απομονωμένο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα στρατηγικό διάλογο με, την, με το Ευρωπαϊκό Αυτοσυμβούλιο. Η κυρία Ράγκελ έθεσε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο Ράγκελ λοιπόν έθεσε το θέμα των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για ορισμένες χώρες, σαν παράδειγμα τη ζώνη ευρώ ή το θέμα της ενισχυμένης συνεργασίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κρατών που δεν ανήκουν στην ομάδα αυτή των κρατών. Το θέμα τίθεται εδώ και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η, συνέλευση δεν έθεσε το θέμα αυτό ουσιαστικά ούτε για το Συμβούλιο ούτε το Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Βέβαια δεν είναι επίγον το θέμα αυτό σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Τι γίνεται με τη συμμετοχή ας πούμε βουλευτών από χώρε οι οποίες δεν μετέχουν ε, στις διαδικασίες ε, για συγκεκριμένα θέματα. Τώρα για τον ρόλο των κοινοβουλευτικών υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα θα έλεγα και άκουσα την έκκληση για επιφυλακτικότητα του Άντριου Ντάφ. Θα ήθελα να πω το εξή Καταρχάς, οργανώσαμε με την κοινή πρωτοβουλία της Πολωνικής Προεδρίας και της Επιτροπής προπολογισμών μια μήνυ συνέλευση, η οποία κράτησε δύο ημέρες, τον Οκτώβριο, και η οποία κατάφερε όπως οι μεγάλες παλιές δύο συνελεύσεις από τη μία να συγκεντρώσει όλα τα ευρωπαϊκά όργανα μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών με 80 βουλευτές από τις χώρες μέλη Κάτι το οποίο επέτρεψε σε κάθε χώρα να αντιπροσωπευθεί με το βασικό κυβερνητικό κόμμα και με την αξιωματική του αντιπολίτευση. Και για δύο ολόκληρες μέρες συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμουμε τους ρόλους ανάμεσα στο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και στους εθνικούς προϋπολογισμούς για να χρηματοδοτήσουμε τη στρατηγική 2020. Η διάσκεψη αυτή πήγε πολύ καλά. Πήγε τόσο καλά που στο τέλος ο εκπρόσωπος της μελλοντική προεδρίας της Δανικής είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτού του είδους η συνάντηση. Προφανώς ένα τόσο τεράστιο θέμα μέσα σε δύο μέρες δεν εξαντλείται και γι' αυτό θα υπάρξει και μια νέα τέτοιου είδους συνάντηση κατά τη διάρκεια του επομένου εξαμήνου. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι ακριβώς το θέμα, αν θα είναι η συζήτηση πάνω στο ίδιο θέμα ή θα υπάρξουν και άλλα θέματα ανάλογα με το χρόνο. Πάντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με εκπροσώπους των κοινοβουλίων και με τους υπουργούς των κρατών μελών ταυτόχρονα. Και αυτό που ήταν το περίεργο είναι ότι η Πολωνική Προεδρία είχε το θάρρος να οργανώσει αυτή τη διάσκεψη, ενώ οι κυβερνήσεις των υπολείπων χωρών και οι υπουργοί τους οικονομικών ήταν κατά. Γιατί οι υπουργοί οικονομικών δεν θέλουν να εκφράζονται μπροστά στους βουλευτές τους, τους εθνικούς, για τέτοιου είδους θέματα. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκαν και ήρθαν. Και έτσι ακούσαμε παράπονα από ορισμένου βουλευτέ, οι οποίοι μάλιστα πολλοί βουλευτέ από τα κράτη-μέλη εκφράστηκαν με διαφορετικό τρόπο από του υπουργού του. Έμοιαζε λοιπόν με τη συνέλευση αυτό που κάναμε. Βέβαια για δύο μόνον ημέρες ήταν μια πρώτη δόση θα έλεγα. Ήταν μια εικόνα έτσι λίγο θολή θα έλεγα του τι μπορεί να είναι μια συνέλευση. Αλλά πάντως αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια γόνιμη αλχημία όπως ε, και στην περίοδο της ε, συνέλευσης μπορούμε να την αναβιώσουμε για να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε τις συνθήκες. Και επανέρχομαι σε αυτά τα οποία είπε στην άλφο θεύνα Αυτό λοιπόν το οποίο όμως με ενοχλεί στα πλαίσια των αναφορών που έχουν γίνει για μια πιθανή νέα συνθήκη, για μια μεταρρυθμιστική συνθήκη, είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα στο εσωτερικό μιας οξυμένης οικονομικής κρίσης και ο ασθενής έχει, άνω των, έχει υψηλό πυρετό άνω των 40. Από τις 27 χώρες, 22 και 23, κάθε πρωί κοιτούν οι ηγέτες του ε, ε, με τι επιτόκια παίζουν το κεφάλι τους. Υπάρχει μια χώρα μέλος η οποία είναι σε, ε, σχεδόν σε πτώχευση και κάποιες άλλες που δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Όσο βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την οξυμένη κατάσταση, το να αφήνει κανείς να, να εννοηθεί, έστω και έμεσα, ότι η λύση, η θαυματουργή είναι η νέα συνθήκη, είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πολλές, ε, ε, πολλές φρούδες προσδοκίες και ταυτόχρονα θα κλονίσει τις αγορές. Ε, τίποτα δεν θα ρυθμίσει πρόθεσμα Σε 10 χρόνια ίσως η μεταρρύθμιση της συνθήκης. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε μπροστά μας είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ότι είναι στην ουσία ένα μέσο το οποίο αν χρησιμοποιήσουμε σωστά μπορούμε να λύσουμε κάποια από τα σημερινά προβλήματα με κάποιες ρυθμίσεις επιμέρους τεχνικές στην υπάρχουσα συνθήκη. Ε, συμπληρωματικά αυτό που ήθελα να πω για τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Πράγματι, στα πλαίσια της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, την οποία συντάσσει η κυρία Μπερές και η οποία θα υποβληθεί στην Ολομέλεια τον επόμενο μήνα και έρχομαι εδώ σε αυτά που έλεγε ο κύριος Γκουερέρο για τη συνάντηση των συντονιστών για το συγκεκριμένο θέμα, θα προταθεί ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τον μήνα Φεβρουάριο κατέτος να γίνεται μια διακοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπροσωπείται ανάλογα με τα θέματα στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, από τις Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων Απασχόλησης και Προϋπολογισμών. Θα πρέπει λοιπόν η πρόταση αυτή, η οποία θα υποβληθεί στην Ολομέλεια, να τύχει της ε, χρήζουσας προσοχής και να προσπαθήσουμε να δούμε αν θα υπάρξει πράγματι δυνατότητα διεύρυνσης των διαδικασιών αυτών και σε άλλα θέματα. Ένας άλλος συνάδελφος, ο ε, Πολωνός Αντιπρόεδρος, του οποίου δεν μπορώ να προφέρω το όνομα, δεν τολμώ φοβάται ότι αν ξεκινήσει η συζήτηση ε, σε σχέση με το θέμα της ε, εγκατάλειψης της ε, κυριαρχίας είναι κάτι που θα ανησυχήσει τους πολίτες βεβαίως. Αλλά αν αφήσουμε εμείς να ξεκινήσει η συζήτηση για μια συνθήκη χωρίς να ορίσουμε το θέμα αυτό τότε θα λέμε ψέματα στους πολίτες. Μια νέα συνθήκη με μια νέα συνέλευση θέλει 5-10 χρόνια. Θα απογοητευτεί ο κόσμος. Είναι τεράστια ιστορία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να εμπλέξουμε τον κόσμο σωστά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πέσει ο πυρετό, θα ξεκινήσει μια συζήτηση. Αλλά να διευκρινίσουμε ότι η συζήτηση αυτή θα κρατήσει πολύ καιρό και δεν είναι μια συζήτηση η οποία είναι πανάκια για τα υπάρχοντα σήμερα προβλήματα. Αυτά λοιπόν συνάδελφοι. Τώρα πρακτικά συμπεράσματα με βάση όλα αυτά. Εγώ μέχρι τώρα έχω διατυπώσει ένα απλό κείμενο εργασίας. Σας προτείνω κύριε Πρόεδρε να υποβληθεί σε μια επόμενη συνάντηση των συντονιστών το εξής ερώτημα. Αν τα θέματα που περιλαμβάνονται στο κείμενο αυτό αξίζουν μια εκθέσεως πρωτοβουλία ή όχι. Και αν τα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό και τα οποία ανέφερα προφορικά και τα οποία συζητήθηκαν πολύ σήμερα σαν παράδειγμα το τι θέση θα πάρουμε απέναντι στη συζήτηση για τη νέα συνθήκη. Υπάρχει ένα θέμα, αυτό το οποίο υπάρχει στο κείμενο εργασίας, για το πώς θα προσαρμόσουμε και θα ρυθμίσουμε τη συνθήκη μέσω ενός gentleman agreement για να βελτιώσουμε καλύτερα την σχέση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον Πρόεδρο το Συμβούλιο Υπουργών και τα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών. Στα πλαίσια της υπάρχουσας συνθήκης επίσης υπάρχει ένα δεύτερο σημαντικό θέμα πάνω στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε εφόσον θέλουμε να παρέμβουμε χρήσιμα, αλλά εδώ απαιτείται μια άλλη έκθεση και φυσικά δεν είμαι υποψήφιος για όλες τις εκθέσεις, Πρόεδρε. Πάντως νομίζω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να τεθεί στους συντονιστές. Καλώς ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λαμασούρ. Εγώ δέχομαι την πρότασή σας να βάλουμε στην υπερήσια διάταξη των συντονιστών στην επόμενη συνάντηση το θέμα. Είναι ένα θέμα σημαντικό, είναι ένα θέμα ευρύ και σαφώς θα πρέπει να μην το αγνοήσουμε. Εντάξει. Περνάμε στο τελευταίο θέμα τώρα στην ημερήσια διάταξη. Πριν περάσουμε στο τελευταίο πρέπει να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Ο κύριος Μάρτιν μας είπε, γιατί δεν μπόρεσε να έρθει, ότι σχετικά με την ακρόαση της Προεδρίας και του Συμβουλίου, την οποία πιστεύαμε να κάνουμε στις 20 Δεκεμβρίου, από πλευράς του δεν υπάρχουν εμπόδια ε, για να γίνει τον Ιανουάριο, 25 Ιανουαρίου. Ε, αυτό κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο προτιμάτε. Δεν ξέρω, ο κύριος ε, Μέντες Δεβίγκο, μπορείτε να μου πείτε αν συμφωνείτε η συνάντηση αυτή να γίνει τον Ιανουάριο. έτσι ώστε η, ακρόαση με το Συμβούλιο να γίνει το Γενάρη για την έκθεσή του και όχι το Δεκέμβριο. Ο Μάρτιν λέει ότι δεν τον ενοχλεί αυτό, οπότε νομίζω ότι συνολικά μπορούμε να είμαστε υπέρ της μετακίνησης τον μήνα Ιανουάριο της συγκεκριμένη συνάντησης με το Συμβούλιο. Κύριος Γκερέρο, συμφωνείτε, διαφωνείτε. Όχι, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Μάρτιν συμφώνησε, όπως είπε ο πρόεδρος. Sì, Μάρτιν ha fatto Μάρτιν. Ο κύριος Μάρτιν, τι λέει. Ο κύριος Μάρτιν που αποσιάσει λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει. E così resta Eh, Περνάμε τώρα στη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Είναι μια κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Εσωτερικών Ελευθεριών για ένα θέμα διαπραγμάτευσης και γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους φίλους που δεν έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στη συνάντηση να φύγουν από την αίθουσα. Θα είναι μια πάρα πολύ συνάντηση γιατί οι διαρμηνείς είπαν ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 12.30. Χαιρετίζω εδώ τους συναδέλφους της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Πρέπει να είμαστε, όπως είπα, πάρα πολύ συνθετικοί.